Uh, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Περίμενα το ανησυχητή και σκιώδη εισηγητές για το πρώτο θέμα της πρωινής ημερήσιας διάταξης που είναι το πρόγραμμα LIFE. Τελικά έχουν καταφτάσει οι αρμόδιοι, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση αυτή για το πρόγραμμα για την ε, δράση για το περιβάλλον και το κλίμα. Το θέμα του Life δηλαδή. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκερμπράντι, τον εισηγητή μας πρώτα απ' όλα το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερος που θα σας παρουσιάσω εδώ το πρόγραμμα live. Είναι η αγάπη μου το πρόγραμμα LIFE είναι το πιο επιτυχημένο, αποτελεσματικό και αποδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λατρεύω. Είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο και είμαι πανευτυχής που ανέλαβα την έκθεση για το πρόγραμμα αυτό. Και χρειάστηκε ακριβώ γι' αυτό να σηκωθώ 5,5 ώρα, άγρια χαράματα για να είμαι στην ώρα μου εδώ. Γιατί λατρεύω ακριβώ αυτό το πρόγραμμα. Και γιατί είναι τόσο μεγαλειώδε. Γιατί τα σχέδια που χρηματοδοτεί είναι καταπληκτικά, έχουν τεράστια προστιθέμενη αξία, ελάχιστα προβλήματα. Πανέμορφο το πρόγραμμα Live. Και εδώ δύο παραδείγματα της τελευταίας διετίας που αποδεικνύουν την επιτυχία του προγράμματο αυτού. Πρόκειται καταρχήν για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε στην Ισπανία, ένα σχέδιο ε, σε ό,τι αφορά τη δηλητηρίαση των ορνίων και άλλων ε, πτηνών, γερακιών και άλλων πτηνών. 600.000 ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα εκατομμύριο από την Ισπανία χρηματοδότησαν ε, την προσπάθεια για να αποφευθεί δηλητηρίαση αυτών των καταπληκτικών αγριοπτηνών. Ε, και δείχνει πως ακόμη και ένα πρόγραμμα με ισχνό προϋπολογισμό μπορεί να έχει τέτοια επιτυχία. Επίσης, ε, στην Ουαλία χρηματοδοτήθηκε ένα σχέδιο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και να δούμε πώς το μεθάνιο από γειτονικέ χωματερές μπορεί να, δεσ... να το δεσμεύσουμε και να το αξιοποιήσουμε οικονομικά. Και αυτό ήταν πολύ επιτυχιασμένα. 1,4 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δημιουργήσαμε ένα πολύ επιτυχημένο σχέδιο και 15.000 λίρε θελήν στον χρόνο μπορούν να χρησιμοποιηθεί από την αξιοποίηση μεθανίου από τι ε, κοντινέ χωματερέ. Και περίπου 30 εκατομμύρια ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε με τέτοια ευγενή προγράμματα και προσπάθειες. Δύο λοιπόν παραδείγματα που αποδεικνύουν το θρίαμβο του life. Είδατε ότι για την έκθεσή μου έχω συντάξει κάποιε τροπολογίε. Μερικές είναι πιο τεχνικού χαρακτήρα, διευκρινίζουν κάπως το κείμενο. Για παράδειγμα, εκεί που λέμε με λίγο άνθρακα, ε, χαμηλό άνθρακα, λέω χαμηλές εκπομπές. Επίσης, εκεί που λέμε διοξίδιο του άνθρακα, λέω αέρια του θερμοκηπίου, γιατί δεν είναι μόνο το διοξίδιο του άνθρακα, έχουμε και το μεθάνιο. Οπότε το αέριο του θερμοκηπίου καλύπτει καλύτερα το θέμα. Και έχω και κάποιες τροπολογίες πιο πολιτικής φύσης. Εκεί που λέμε καθαρή ενέργεια, αναφέρω τι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Επίσης, εκεί που λέω τα θαλάσσια ενδιατήματα είπα γενικά οικοσυστήματα ή ενδιατήματα Γιατί δεν μιλούμε μόνο για τη ε, βιοπικιλότητα στα θαλάσσια ε, οικοσυστήματα, γιατί και τα χερσαία ενδιατήματα είναι εξίσου σημαντικά. Επίση τόνισα τη σημασία που έχει η, η σωστή αξιοποίηση των πόρων και επίσης ε, αναφέρω και την κυκλική οικονομία. Θα ήθελα να σταθώ τώρα σε καμιά δυο τροπολογίες που είναι πολιτικού χαρακτήρα, μείζωνος πολιτικής σημασίας. Καταρχήν ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος και θα παραμείνει περιορισμένος ε, Εκτό και προτείνουμε αύξηση. Εγώ προτείνω από 5,4 δι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανέλθει σε 7,2 δισεκατομμύρια ο προπολογισμό του ΛΑΙΦ, κάτι που ευθυγραμμίζεται με προηγούμενε ε, θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ του ΛΑΙΦ. Και προσβλέπω στη δική σα υποστήριξη για να περάσει η πρόταση για την αύξηση του προπολογισμού. Επίση, και πάλι σε σχέση με προηγούμενε δηλώσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, για, το, για τη συμπερίληψη του περιβάλλοντος προτιμούμε από 25% σε 30% να περάσουμε ε, στη συνεκτίμηση του περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά τώρα το συντελεστή χρηματοδοτηση άλλο σημαντικό θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε κάποια ελαστικότητα στη θέσπιση του ποσοστού του συντελεστή χρηματοδότηση. Δεν είμαι κατά αλλά στι τροπολογίε μου προσπάθησα να μην προσδιορίζω τον ακριβή συντελεστή, αλλά τις προϋποθέσεις για το ελάχιστο και το ανώτατο όριο σε χρηματοδότηση. Και θα το βρείτε αυτό και πάλι στι τροπολογίε. Άλλο σημαντικό στοιχείο που επίσης ε, έχει πολιτική διάσταση είναι η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματο. Η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε ε, κάτι ε, ανεπαρκές κατά τη γνώμη μου. Εμείς θέλουμε μια ουσιαστική διάμεση αξιολόγηση μετά από μια τριετία και όχι από, μετά από μια τετραετία όπω προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπω και κάποια κριτήρια στι τροπολογίε για να εξασφαλιστεί μια ποιοτική διάμεση αξιολόγηση που θα δράζεται στις επιδόσεις, στα αποτελέσματα. Και επίσης το θέμα δεν είναι η αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση καθ' αυτή αλλά ποια στοιχεία θα προκύψουν, ποια δεδομένα θα προκύψουν από μια αξιολόγηση και θα πρέπει να ληφθούν όντω υπόψη. Άλλο σημαντικό θέμα είναι τα αναξιοποίητα κονδύλια του τρέχοντος προγράμματος LIFE. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί να μεταφερθεί στο πρόγραμμα Invest. Εγώ θα προτιμούσα να επιστρέψουν στο νέο πρόγραμμα LIFE θα χρησιμοποιεί τα κονδύλια. Γιατί σίγουρα οι περιβαλλοντικέ επιδόσεις του LIFE είναι πολύ ανώτερε από τι περιβαλλοντικέ επιδόσεις του EU Invest, που είναι γνωστό ω το Ταμείο Juncker. Οπότε και αυτή η τροπολογία είναι σημαντική. Άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη μου έχει κρίσιμη σημασία και είναι κάπως ακαθόδες στη συζήτηση με τα κράτη-μέλη, δεν θα ήθελα τα κονδύλια του LIFE να υποκαταστήσουν ε, εθνικά κονδύλια. Γιατί τα τελευταία 5 με 10 χρόνια είδαμε ότι οι δαπάνες για τη βιοπικιλότητα στα κράτη-μέλη έχει μειωθεί αισθητά και πολλά κράτη-μέλη προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις εθνικές τους δαπάνες χρησιμοποιώντας κοινοτικά κονδύλια. Αυτό κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνη τάση, γιατί χρειαζόμαστε ε, τα ψηλά κονδύλια παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλότητα και δεν θα πρέπει να αντικαθιστούμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς με το κοινοτικό προϋπολογισμό γιατί το, το Συμβούλιο πολύ θα ήθελε να εφηγραμμίσει το LIFE με τα εθνικά προγράμματα βιοπικιλότητας και από άποψη πολιτικής δεν έχω πρόβλημα αλλά από δημοσιονομική άποψη διαφωνώ. Και τα τελευταία δύο στοιχεία στην πολιτική συζήτηση που είχαμε για το προηγούμενο και για τα προηγούμενα προγράμματα live ε, ε, για το θέμα των εθνικών ε, κονδύλιων και την κατανομή των εθνικών κονδύλιων. Εγώ πιστεύω ότι το live θα πρέπει να παραμείνει τόσο επιτυχημένο και προσανατολισμένο στα αποτελέσματα όπως τώρα. Θα πρέπει δηλαδή η ποιότητα να είναι το ζητούμενο και όχι η ειδική γεωγραφική κατανομή. Δηλαδή θα πρέπει εκ των προτέρων να κάνουμε μία κατανομή μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί έτσι δεν θα χρηματοδοτούνται χρήματα αλλά προς τα σχέδια, αλλά τα σχέδια θα απορροφούν χρήματα. Δεν είναι, είναι προθύστερο, είναι λάθος σχήμα αυτό. Μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Το Κοινοβούλιο θέλει και πάλι εθνική κατανομή. Είμαι έτοιμος να το συζητήσω με το Συμβούλιο αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εμείνουμε στην ανάγκη ποιότητας και από επιδόσεων και να βρούμε μια λύση με το Συμβούλιο. Τέλος, το πρόγραμμα LIFE έχει ένα διόλο μελιτέο προϋπολογισμό, 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρό ποσό, και ένα πολίτη πραγματικά θα εντυπωσιαστεί. Αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό πραγματικά και αυτό το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα τέτοιο μεγάλο επίβολο πρόγραμμα. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει στην πρότασή τη ότι το LIFE ε, μπορεί να αποδώσει με τόσο μικρό προπολογισμό αν επιτύχουμε ε, στην ανάγκη συνεκτίμησης ε, των κλιματικών αλλαγών του περιβάλλοντος, της κυκλικής οικονομίας, τα μεγάλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της πολιτικής συνοχής και της κοινή γεωρικής πολιτικής. Θα πρέπει και εκεί να συνεκτιμούνται αυτές οι διαστάσεις και αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση μπορούμε να αρκεστούμε σε ένα σχετικά περιορισμένο προϋπολογισμό αν έχουμε στα μεγάλα προγράμματα δαπανών συνεκτίμηση των διαστάσεων περιβάλλοντος κλιματικών αλλαγών και κυκλικής οικονομίας στα άλλα βασικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το LIFE δεν μας δίνει εχέγγυα επιτυχίας. Γιατί και στη Γεωργία και στη Συνοχή τα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να καταργήσουν ε, την περιβαλλοντική αιρεσιμότητα και μερικές φορές και από το Κοινοβούλιο ξεκινούν τέτοιες φωνές. Οπότε εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ένα είδος αξιολόγησης μετά τη λήψη της απόφασης και μετά τη συμφωνία με το Συμβούλιο επί του συνόλου των δαπανών του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου να γίνει κάποιο είδος αξιολόγηση και να δούμε ε, τι ποσοστό επιτυχίας έχει το mainstreaming. Γιατί αν συνεκτιμάτε, αν δεν συνεκτιμάται παρκώς το περιβάλλον ε, στα άλλα προγράμματα, θα πρέπει να αντιδράσουμε για να το διορθώσουμε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο βέβαια. Και συζητώ με τους και οδησηγητές, με την ε, Επιτροπή και με άλλους για να δούμε πώς θα το εξασφαλίσουμε. Μία επαρκή συνεκτίμηση ε, των περιβαλλοντικών ε, κριτηρίων και στις άλλες μεγάλες δαπάνες. Δεν θα πρέπει οι περιβαλλοντικές δαπάνες να περιορίζονται μόνο στο πρόγραμμα LIFE, ενώ στη, στα μεγαλεπίβολα προγράμματα με τους ε, παχυλούς προϋπολογισμούς, όπως είναι η συνοχή και η κοινή γεωρική πολιτική, να μην πλήρουν αυτούς τους περιβαλλοντικούς στόχους. Γιατί κάτι τέτοιο θα αποδυναμώσει και το LIFE και θα μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τους στόχους. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδης ηγητές για τη μέχρι τώρα συνεργασία και να πω ότι ανυπομονώ για τη συζήτηση και εδώ στην Επιτροπή Έμβη και προσβλέπω σε μια πολύ θετική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα LIFE. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το ΕΛΚΑ η κυρία Γιούσο που εκπροσωπεί τον ε, Σκιώδη Ντόντα. Καλημέρα σας. Ο κύριος Νταντά ε, μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω. Από πλευράς του κυρίου Νταντά να σας διαβάσω το Ευχαριστώ τον συνάδελφο Γκέμπραντι για την εργασία του και για την ε, διαβούλευση που έκανε με όλους πριν υποβάλει τις τροπολογίες. Η έκθεση του κυρίου Γερμπράντη προτείνει πολλές αλλαγές τις οποίες στηρίζω ο επανακαθορισμός της χρηματοδότησης των υποκατηγοριών. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να στηρίξουμε την ε, μετάβαση της γεωργίας προς πιο βιώσιμες πρακτικές. Και γι' αυτό προτείνω να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο ε, αποκαλώ ε, πρόγραμμα για ε, βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, το οποίο περιλαμβάνει και τη χρήση των υπολείπων υδάτων. Πρέπει επίσης να, λαμβάνει πάντα υπόψη, να λαμβάνουμε πάντα υπόψη στην γεωργία και την ενέργεια την περιβαλλοντική πλευρά. Γι' αυτό τονίζω ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτεί το life δεν θα πρέπει να αμφισβητούν τις προτεραιότητες άλλων νομοθετημάτων της Ένωσης. Επίσης θα επαγρυπνήσω για να συμμετάσχει συγκεκριμένα η κοινωνία των πολιτών και οι διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες, ούτως ώστε το πρόγραμμα αυτό να είναι ε, κοντά στην επίλυση των ε, προβλημάτων των πολιτών. Επίσης, θα πρέπει και τρίτες χώρες να είναι επιλέξιμες και ενδεχομένως και υποψήφιες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τους όρους βάσει των οποίων νομικά πρόσωμα σε τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν, ιδίως ε, συνδεδεμένες. Επίσης, ο εισηγητής θα πρέπει να λάβει υπόψη τις άκρος ε, περιφερειακές περιοχές και τις υπερπόντιες ε, περιφέρειες και εδάφη. Ιδίω αυτές που είναι ε, μακριά από οποιαδήποτε άλλη ξηρά. Η πρωτοβουλία BEST από το 2011 μας έχει κάνει να καταλάβουμε την οικολογική σημασία των ε, άκρος περιφερειακών περιοχών και των υπερποντίων εδαφών για την εγγύηση της βιοποικιλότητας. Η έκθεση λοιπόν πρέπει να διατηρήσει την επιλεξιμότητα αυτών των ε, εδαφών για τα προγράμματα live. Αυτά ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χερμπράντη για την ε, πολύ καλή έκθεση η οποία καλύπτει και πολλές από τις δικές μου παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των τεχνικών συνεδριάσεών μας, που ήταν πολύ επικοδομητικές. Τον ευχαριστώ πραγματικά για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε με όλους εμάς τους σκιώδης εισηγητές. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία απασχόλησης. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να το πούμε με τρόπο στεναρό και θα το πει ελπίζω και η Επιτροπή Άγκρη με τη γνωμοδότηση που ετοιμάζει ε, απέναντίας για την ευημερία, την κοινωνική και την οικονομική μακροπρόθεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να αποφύγουμε την αποδυνάμωση της βιοπικιλότητας και να φροντίσουμε να υπάρξει η μετάβαση στην κυκλική οικονομία και η απαλλαγή μας από τον άνθρακα. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει να ε, σταθώ σε ορισμένα σημεία για να βελτιωθεί η πρόταση κανονισμού για το live. Θα υποβάλω βεβαίως τις σχετικές τροπολογίες. Διότι ασχολούμαστε και με μια ομάδα εργασίας του Κοινοβουλίου ε, με το πρόγραμμα live ούτως ή άλλως και θα δω τα πορισμένα θα προκύψουν και από εκεί. Πάντω πρέπει να αυξήσουμε την ε, ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα αυτό σε μια πρώτη φάση, ακόμα και με μια επικοινωνιακή στρατηγική που να είναι πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική και να διοχετευτεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Το live και η ενέργεια από ορυκτά καύσιμα. Έχει να κάνει με την καύση ορυκτών καυσίμων για τις μεταφορές, την θέρμανση και για τα κλιματιστικά η απαλλαγή από τον άνθρακα στους τομείς αυτούς ε, έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα του της ατμόσφαιρας και στην υγεία των πολιτών. Θα πρέπει να, να αναζητήσουμε νέες πηγές ενέργειας και το πρόγραμμα LIFE θα επιτρέψει να χρηματοδοτηθεί ή ο εξοπλισμός των νοικοκυριών με καλύτερα μηχανήματα που να μην βασίζονται πλέον στα ορυκτά καύσιμα και να επιτρέψουν την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τρίτο σημείο, όπως είπε και ο συνάδελφος Χερμπράντη, για το πρόγραμμα LIFE η ενδιάμεση αξιολόγηση θα είναι ένα πρώτο, ε, μια πρώτη συνολική εικόνα του πώς πήγαν οι αλλαγές που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν. Χρειάζεται πραγματική εξωτερική και ανεξάρτητη αξιολόγηση η οποία να προσφέρει λογικές εύλογες εγγύησεις για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και προκειμένου να επιδιώξουμε τις περιβαλλοντικές μας φιλοδοξίες. Είναι καθοριστική σημασία να πάρουμε τις πρωτογενείς χρηματοδοτήσεις ε, για το πρόγραμμα του προγράμματος LIFE για την προστασία του περιβάλλοντος, την ε, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την προσφορά καθαρότερης ενέργειας στους πολίτες. Είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να, να γίνουν πιο υπεύθυνε για όλες τις πτυχές που αφορούν το περιβάλλον και να αλλάξουν τι πρακτικέ του για να δημιουργούν το δυνατόν λιγότερη πίεση και ζημιέ στο περιβάλλον. Αυτή η ανανεωμένη ευθύνη του κόσμου των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ένα, σημείο, ένα στοιχείο κλειδί στι στρατηγικέ του προγράμματο LIFE για να επιδιώξουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι, χρηματο... οι ιδιωτικέ χρηματοδοτήσει, του ιδιωτικού δηλαδή τομέα, θα επιτρέψουν να ε, προχωρήσουν προγράμματα που πολλέ φορέ απλώ δεν ε, προχωρούν λόγω έλλειψη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στα ε, προγράμματα του LIFE, τα οποία μπορούν να επαναληφθούν και να μεταφερθούν και αλλού, για να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθηθούν προγράμματα τα οποία μπορούν να λάβουν επενδύσει και που μπορούν οικονομικά να είναι βιώσιμα. Επίση, δύο παρατηρήσει για του ολοκληρωμένου στόχου. Πρώτον, δεν είναι ίση η κατανομή των κονδυλίων live στα κράτη-μέλη. Και οι εθνικές αρχές δεν είναι αποτελεσματικές στο να εγγυηθούν την πιο ισόρροπη εκτέλεση των ίδιων των προγραμμάτων. Η επιλογή των προγραμμάτων βάσει της, ε, της αξίας τους, του περιεχομένου τους, θα πρέπει να οδηγήσει και σε πιο ισότιμη κατανομή των κονδυλίων για να υπάρχει αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των προγραμμάτων live στα κρατημέλη και αυτά να φροντίζουν, δηλαδή τα κρατημέλη να φροντίζουν να προτείνουν ποιοτικότερα προγράμματα με καλύτερη γεωγραφική ισορροπία. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται και από τη συμπληρωματική, την επιπλέον χρηματοδότηση που θα βρούμε. Μέσω κυρίω του συνδυασμού του περιβάλλοντο με το κλίμα σε όλε τι βασικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω την ΚΑΠ και την πολιτική συνοχή. Είναι και τα δικά του εργαλεία χρηματοδότηση. Ε, Παρατηρώ ότι τα σημεία επαφή του προγράμματο LIFE ε, χρειάζεται να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο για να υπάρχει αυτή η ελάχιστη παροχή υπηρεσιών στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια. Και επίση πρέπει να παρακολουθήσουμε πώ λειτουργούν και να υπάρχουν ε, και εκθέσεις για το πώ λειτουργούν με ε, δείκτε συγκριτική αξιολόγηση και ποιοτικού δείκτε. Και να εξετάζουμε προσεκτικά τι δυνατότητε μείωση του κόστου ώστε ε, να έχουμε σωστή ε, καταγραφή του κόστους ωφελίας ε, και της βελτίωσης των προγραμμάτων LIFE. Από τη δική μου τη σκοπιά πρέπει να εγγυηθούμε την συμπληρωματικότητα του LIFE με άλλα κονδύλια και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην υπάρχουν επικαλύψεις με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το τόσο σημαντικό πρόγραμμα. Εν τέλει, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του ίδιου του LIFE, θεωρώ ότι η πρικοδότησή του για την υλοποίηση θα πρέπει ε, να αυξηθεί. Είναι τελείως ανεπαρκής αυτή τη στιγμή, όπως θα παρατηρήσει ε, φαντάζομαι και το Κοινοβουλίο. Ε, χρειάζονται περισσότερα κονδύλια πρέπει να προβλεφθούν γιατί είναι σημαντικό. Για το πρόγραμμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, να δείξει ότι έχει πολύ ε, υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ορισμένη σκιώδηση είναι απόνδεση. Υπάρχει χρόνος. Γι' αυτό επέτρεψα στον κύριο Καπούτο ε, όσο χρόνο ήθελα να παρακαλώ τους επόμενους ομιλητές να σέβονται το χρόνο. Δεν βλέπω κανένα σκιώδη. Δεν ξέρω αν τον αντικαθιστά κανείς. Αν όχι, για τους πράσινους θα μιλήσω εγώ. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δώσω το καλό παράδειγμα να μιλήσω σύντομα. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Γερμπράντη και την Επιτροπή για το έργο τους. Πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι καλή βάση για περαιτέρω εργασία, όπως και το σχέδιο εκθέσεις Που είναι πολλά υποσχόμενο. Αλλά ο χρόνος είναι λίγος. Άρα πρέπει να καταλήξουμε στα βασικά στοιχεία με επαρκείς λεπτομέρειες για κάποια σημεία που ανέφερε και ο εισηγητής, ε, ο προϋπολογισμός, η χρηματοδότηση, οι δείκτες, συνέπεια με άλλες ενωσιακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένες της κοινή γεωργικής πολιτικής κλπ. Λοιπόν, κάποια άλλα σημεία που για τους πρασίνους είναι σημαντικά και τα οποία θα εκφραστούν και μέσω των τροπολογιών μου. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, μείωση της ε, βιοποικιλότητας και οι χώροι Natura 2000 να χρηματοδοτηθούν επαρκώς. Στηρίζω τον εισηγητή να αυξηθούν οι πόροι λοιπόν για το live, αλλά πρέπει να δούμε και πέρα από το πρόγραμμα Πρέπει η βιοπικιλότητα να περιέχεται σε όλα τα πρόγραμμα και να μπορούμε να την εντοπίζουμε σε όλα τα ενωσιακά προγράμματα. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το παρόν θέμα, αλλά να το έχουμε υπόψη. Δεύτερον, καλύτερη διακυβέρνηση, συμμετοχή του κοινού, διαφάνεια, καλύτερη επικοινωνία και οι δυνατών και συμβουλές για ενδεχόμενους δικαιούχους, ε, προσπαθώντας να συμπεριλάβουμε όλες τις περιφέρειες. Κάποιοι δικαιούχοι πρέπει να στηριχθούν για να μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Συμφωνώ με τις κατηγορίες που προτείνει η Επιτροπή, τις κατηγορίες προγραμμάτων, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε και περιθώριο για τη δημιουργία δυναμικού, ιδιαίτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση, και για μικρότερα προγράμματα από ΜΚΙΟ, έτσι είχαμε την πείρα από τα προηγούμενα προγράμματα. Οι τοπικές πρωτοβουλίες και οι μικρές ΜΚΟ ε, δεν μπορούσαν εύκολα να επωφεληθούν από το live. Συμφωνώ με τον κύριο Χεμπράντη, πολύ σωστή και η γεωγραφική ισορροπία. Να φτιάξουμε ένα σύστημα που να βασίζεται στα φυσικά χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις, ε, τους βιογεωγραφικούς ε, προσδιορισμούς. Έχουμε τέτοιους ε, προσδιορισμούς και διαχωρισμούς στην Ευρώπη και όχι απλώς τα κρατικά σύνορα. Από μια οικολογική πλευρά τα πολιτικά σύνορα δεν έχουν έννοια. Τέλος, καλύτερη επίβλεψη επίσης. Εξάντε και εξπόστα αξιολόγηση και για τα προγράμματα αλλά και για να υπάρχουν ε, δικλείδες ασφάλειας, ούτως ώστε τα προγράμματα αυτά να μην ε, ακυρώνονται από άλλα ενωσιακά προγράμματα. Όπως είπα γενικά είναι πολύ θετική η γνώμη μου, μπορούμε να εργαστούμε επικοδομητικά για να βρούμε κοινό τόπο με τους συναδέλφους και να στείλουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ ότι το LIFE είναι πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ουσιοδός το πρόγραμμα, απλώς να προωθήσουμε περαιτέρω βιώσιμες λύσεις με σωστό και διαφανή τρόπο και να διασφαλίσουμε πρόσβαση στην χρηματοδότηση για μικρότερους φορείς όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι μικρές μη κάπα ελπίζω να μην υπερεύει το χρόνο μου και τώρα, επόμενο ο για την ΚΟΕ. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω το σκιώδη ούτε του EFTD. Οπότε, παρακαλώ, όποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν τον λόγο. Και, και πρώτη είναι η κυρία Μένιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, υποστηρίζω ότι χαίρομαι που ο κύριος Γκεμπράιντ υπέβαλε αυτή την έκθεση η οποία μου φαίνεται πολύ καλή. Όμως ξέρω τι έγινε στην Άγκρη. Έκαναν διάφορα περίεργα υπόγεια πράγματα. Νομίζω ότι εμείς ε, όμως θα πάμε καλύτερα γιατί έχουμε πολύ καλό εισηγητή. Άριστο και τον συγχαίρω. Όπως ξέρετε υπήρξε ένα ψήφισμα στις 14 Μαρτίου στο οποίο καταλήξαμε από κοινού και όπου λέμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι πιστώσεις για το πρόγραμμα. Αναφερθήκαμε τώρα στη βιοπικιλότητα, κυκλική οικονομία, ενεργειακή μετάβαση. Όλα αυτά στις επόμενες δεκαετίες και αιώνες θα καθορίσουν τη ζωή μας. Άρα χρειαζόμαστε και περισσότερο χρήμα. Αλλά ο κύριος Γκεμπράντη έχει δίκιο. Φυσικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Ιδιαίτερα μέσω της γεωργικής και μέσω της πολιτικής συνοχής για να προωθήσουμε και μέσω αυτών των πολιτικών την περιβαλλοντική πολιτική. Είμαι πολύ κοντά στη σκέψη του λοιπόν και θεωρώ ότι με τον εισηγητή και τους κοιόδης θα τα καταφέρουμε. Να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα από το Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε και την πλειοψηφία, ούτω ώστε το πρόγραμμα LIFE να προωθήσει τους στόχους του. Η ενεργειακή μετάβαση, για παράδειγμα, στη Γερμανία. Εμείς έχουμε ακόμη ενέργεια πολυγνήτη στο κράτος μου στη Γερμανία. Και εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν πράγματα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή η περαιτέρω συζήτησή μας στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μπρέναν. Ευχαριστώ. Έχω τρεις παρατηρήσεις και μία, ερώτηση. Καταρχήν, όταν ε, ε, είχαμε την έκθεση του IPCC και είπαμε ε, ότι έχει νόημα να περάσουμε το 25% στο 30% για τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά όχι... όχι, μάλλον το 25% είναι καλό. Τώρα το 30% δεν ξέρω ε, πώς το τεκμηριώνεται. Και βλέπω το επιχείρημα για τη συνεκτίμηση των κλιματικών αλλαγών. Αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε και αντίθετα. Γιατί το να ζητήσουμε αύξηση του προπολογισμού, πως θα υπονομεύσουμε το επιχείρημα του mainstreaming. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να επιχειρηματολογήσετε. Τώρα το δεύτερο και τρίτο σχόλιο σχετίζονται με το Brexit και συγγνώμη που το θίγω. Ε, ποια είναι η αναλογία του Ηνωμένου Βασιλείου στο live και με το Brexit τι θα γίνει με το χάσμα που θα δημιουργηθεί, με το κενό που θα δημιουργηθεί. Και ένα συναφές τρίτο θέμα. Με το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχει κάποιο σχέδιο για να διατηρηθούν κάποιοι δεσμοί και πέραν του Brexit για να συνεχίσουμε να ε, αξιοποιούμε τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις μας και τα θετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα μιμούμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα Νάπαλη. Αυτό, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, δεν βλέπω να ζητά άλλος κανείς το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ντελγάδο Ρώσας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ θετική αξιολόγηση που κάνετε για το πρόγραμμα LIFE και συμφωνούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το LIFE διαδραματίζει έναν μοναδικό, ιδιαίτερο και πολύ θετικό ρόλο. Και θα ήθελα να απαντήσω στα πολιτικά σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Το πρώτο ζήτημα αφορά τον προϋπολογισμό και την πρόταση που κάνετε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του LIFE. Καταρχήν στη δική μας πρόταση προτείνουμε 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ στα σχέδια για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές που ήδη συνιστά αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο και με επίσης έχουμε 46% αύξηση στις δράσεις για τα περιβαλλοντικά υποπρογράμματα αν τα συγκρίνουμε με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Και πέραν αυτής της αύξησης και δεδομένου του καταλητικού ρόλου που διαδραματίζει το LIFE το ενισχύουμε περαιτέρω. Για παράδειγμα, στα στρατηγικά ολοκληρωμένα σχέδια έχουμε μία ενίσχυση και χρηματοδότηση και από άλλες πηγές. Επίσης, ενισχύονται προγράμματα που περιλαμβάνουν και το σκέλος φύση και επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στη συνεκτίμηση ε, της φύσης και έχουμε και χρηματοδότηση καλύτερη της βιοποικιλότητας. Με όλα αυτά τα επιπλέον μέτρα θα έχουμε μια συνολική αύξηση του LIFE στα περιβαλλοντικά και κλιματικά σχέδια στο επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάτι που είπε ο κύριος Γκερμπράντη και άλλοι είναι ότι δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το δυναμικό που έχει το LIFE να λειτουργήσει ως καταλήτης θα αξιοποιηθεί αν και στους άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς συνεκτιμάται το κλίμα και το περιβάλλον. Ε, και έτσι συμβάλλουν και τα άλλα προγράμματα στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών μας στόχων. Το LIFE δεν είναι μόνο πολιτική, είναι εργαλείο και συμπληρώνει τα υπόλοιπα ταμεία. Και αυτό το χαρακτήρα έχει και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά τα ταμεία θα πρέπει να εξυπηρετούν τις περιβαλλοντικές μας πολιτικές. Φυσικά το LIFE θα πρέπει να συνάδει και με τις άλλες, α, τους άλλους στόχους πολιτικής, αλλά και οι υπόλοιπε πολιτικές θα πρέπει να συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς μας στόχους. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, τα ολοκληρωμένα στρατηγικά προγράμματα για τη φύση, είναι σημαντικά. Συχνά μα είπατε ότι από το Ρατούρα 2000 δεν υπήρχαν αρκετά κονδύλια για τη βιοπικιλότητα. Και ακριβώ προσθέτουμε κριτήρια για να αντλήσουμε περισσότερα κονδύλια και μέσω της συνεκτίμησης των περιβαλλοντικών κριτηρίων, αλλά και κυρίως για να αξιοποιήσουμε πλήρως την πολιτική μας για τη βιοπικιλότητα. σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή και τη γεωγραφική ισορροπία, αυτή τη στιγμή το LIFE δεν ε, χαρακτηρίζεται από γεωγραφική ισορροπία. Θέλουμε να βρούμε λύσεις για αυτό το θέμα. Και συμφωνώ ότι η σωστή προσέγγιση δεν είναι η εθνική, τα εθνικά κονδύλια. Γιατί στο παρελθόν δεν ήταν πολύ θετική η πρόταση αυτή και σίγουρα μόνο ενισχυμένη συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφής θα μας επιτρέψει να διαδώσουμε τους μηχανισμούς και τα εργαλεία παντού στην Ευρώπη για να αυξηθεί η επιτυχία του LIFE. Επίσης, πρόταση για αύξηση από 25% σε 30% του σκέλους για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει οριζόντια θέση για το 25% για το κλίμα. Και αυτό δεν ενοχλεί το LIFE, γιατί όχι μόνο έχουμε ξεχωριστό πρόγραμμα για το κλίμα, αλλά φαντάζομαι ότι σχεδόν σε όλα τα άλλα σχέδια και προγράμματα θα υπάρχει ε, μια συμβολή του ώστε να μετριάσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά και για, το, για τη φύση και τη βιοποικιλότητα τα πλεονεκτήματα φτάνουν μέχρι και το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα και το συντελεστή συγχρηματοδότησης, όντως με την πρότασή μας θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ε, μεταβλητές ε, απαιτήσει για, τα τα επιμέρους προγράμματα και να επικεντρωθούμε και να λάβουμε όψη τι ανάγκε των δικαιούχων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ελαστικότητα, την οποία προβλέπουμε στη νέα πρόταση. Τώρα, αν θεσπίσουμε αύξηση του συντελεστή τη χρηματοδότηση, ε, ή προτείνουμε ένα μέγιστο συντελεστή που είναι σημαντικό για κάποιου δικαιούχου, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο συνολικός αριθμός των χρηματοδοτούμενων σχεδίων θα μειωθεί. Επίσης, αν θα σπίσουμε ένα ελάχιστο συντελεστή συγχρηματοδότηση, αυτό σημαίνει ότι κάποια σχέδια θα πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συντελεστή ίσω υψηλότερο από αυτό που θα πρότειναν ή θα χρειάζονταν κάποιοι ετούντε. Γι' αυτό εμεί προτιμούμε να διαφυλάξουμε μια ευελιξία και ελαστικότητα. Τώρα το θέμα της αξιολόγησης του LIFE και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αναγνωρισμένη μέχρι στιγμής επιτυχία του LIFE προέρχεται και από τις ε, αξιόπιστες αξιολογήσεις που έγιναν. Βέβαια, κάποια προγράμματα live είναι χρονοβόρα και πολυετή. Τα προγράμματα για τη φύση ξεπερνούν την τριετία συνήθως. Οπότε, αν έχουμε μια περίοδο αξιολόγησης, ενδιάμεση αξιολόγησης πριν την τετραετία, δεν θα έχουμε προλάβει να συγκεντρώσουμε κατάλληλα στοιχεία και απαρκή στοιχεία για μια ε, αξιόπιστη αξιολόγηση. Γιατί αν την κάνουμε πολύ πρόωρα την αξιολόγηση, θα πρέπει ε, να πάμε προς το προηγούμενο πρόγραμμα live και να επεκτείνουμε την αξιολόγηση και στην προηγούμενη περίοδο του live. Γι' αυτό και εμείς προτιμούμε την τετραετία για την ενδιάμεση αξιολόγηση και όχι νωρίτερα την τριετία δηλαδή. Και λίγα σχόλια καταληκτικά. Καταρχήν ο ιδιαίτερος λόγος των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των ε, νησιωτικών περιοχών. Όντως, ανοίγουμε το πρόγραμμα ώστε να ανοίξουμε το πρόγραμμα, το προηγούμενο BEST και για τα, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις υπερπόντιες περιοχές. Θέλουμε φυσικά και τρίτες χώρες να μπορούν να επωφεληθούν από το LIFE και γι' αυτό προτείνουμε μία προσέγγιση με δύο φάσεις, κάτι που απλουστεύει τη διαδικασία για την αίτηση επιχορηγήσεων και την πρόσβαση στο live. Βέβαια, υπάρχουν πολλά και διάφορα προγράμματα διαφορετικών, ε, διαφορετικής εμβέλειας, ώστε να προσαρμόζεται στη στις ανάγκες των δικαιούχων. Σε ό,τι αφορά το Brexit και τι θα γίνει στο μέλλον, η πρόσβαση των τρίτων χωρών στο live επιτρέπεται, αν το επιθυμούν φυσικά οι τρίτες χώρε. Και μακάρι το, το Ηνωμένο Βασίλειο, ό,τι και γίνει στο μέλλον, να παραμείνει συνδεδεμένο και να έχει πρόσβαση στο live. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον εισηγητή για τις τελικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. που ασχοληθήκαν τόσο σοβαρά με το θέμα αυτό και την έκθεσή μας. Ελπίζω ότι θα περάσουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία για να ολοκληρώσουμε. Μερικές παρατηρήσεις μετά τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω τον Νίκολα Καπούτο για τη δουλειά του στη δουλειά, στην Επιτροπή Γεωργίας. Και μετά την ψηφοφορία της Τρίτης πρέπει να πω ότι το αποτέλεσμα ίσως δεν θα ήταν τόσο καλό όσο επιθυμούσαμε μεν, αλλά Κοιτάζω πάντοτε με περιέργεια το τι θα συμβεί στην Επιτροπή Γεωργία, διότι το πρόγραμμα LIFE είναι λιγότερο από 1% τη συνολική ε, δυνατότητα του ΚΑΠ και τελικά παίρνουν περισσότερα κονδύλια από το LIFE από ό,τι θα μπορούσαν. Δεν το πολύ καταλαβαίνω, κυρίω γιατί τόσα πολλά δαπανώνται για την κοινή αγροτική πολιτική με τρόπο αναποτελεσματικό και χωρί να έχουμε. Ε, τη σωστή επιδίωξη των στόχων μας να το σκεφτούμε αυτό όταν θα ασχοληθούμε με τη δική μας την έκθεση. Ο κύριος Μπρέναν είχε κάποιες ερωτήσεις για τον εξορθολογισμό. Νομίζω ότι το απάντησε αυτό εν μέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο σκοπός του LIFE είναι να λειτουργήσει καταλυτικά θα έλεγα, δηλαδή να πυροδοτήσει κάποιες αντιδράσεις. Ο εξορθολογισμός είναι ζωτική σημασίας. Εγώ είμαι υπέρ τη λογική του να μην χάσουμε καθαρή αξία στον τομέα τη βιοπικιλότητας. Πιστεύω ότι ούτε οι δαπάνε τη γεωργία, ούτε οι δαπάνε τη συνοχή θα πρέπει να έχουν ε, αρνητικέ συνέπειε για τη βιοπικιλότητα. Αυτό είναι εξορθολογισμό και αυτό θα πρέπει να είναι η βάση των ευρωπαϊκών δαπανών και γενικώ των δημοσίων δαπανών. Φοβούμε ότι Απέχουμε λίγο ακόμη από το στόχο αυτό, αλλά αυτό θα επιδιώξω εγώ. Δεδομένης της πολιτικής πραγματικότητας, σίγουρα ε, υπάρχει μεγάλη πίεση σε μια διψωνακή γραμμή όπως αυτή του live, γιατί ο εξορθολογισμός ίσως τελικά να μην είναι τόσο επιτυχής όσο θα επιθυμούσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη απήντησε στις ερωτήσεις για το κατά πόσον το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον μετά το Brexit θα μπορεί να είναι επιλέξιμο. Να σας παραπέμψω στο άρθρο 11 που μιλά για τους επιλέξιμους φορείς, τα επιλέξιμα πρόσωπα και λέει ότι τις χώρες που συνδέονται με τμήματα του προγράμματος μπορεί να είναι επιλέξιμες. Όλα εξαρτώνται λοιπόν από το πώς θα διαμορφωθεί το Brexit. Θα είναι σκληρό. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει δυσκολία να συνδεθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με το πρόγραμμα και να είναι επιλέξιμο. Είναι ένα σημαντικό λοιπόν στοιχείο, πρέπει να ληφθεί υπόψη στι διαπραγματεύσει για τον Brexit. Εγώ σα παρακαλώ να παραμείνετε συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, για να μπορείτε κι εσεί να υποφεληθείτε από το πρόγραμμα LIFE. Τέλο, Πρόεδρε, ο Νίκολα Καπούτο και άλλοι σκιώδει με ευχαρίστησαν για το πνεύμα συνεργασία που επιδεικνύουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ το βοηθό μου τον Ρόμπερτ. Γιατί έχει δημιουργήσει στις τεχνικές συνεδριάσεις ένα τέτοιο κλίμα που είναι ευχάριστο σε όλους μάλλον. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι οι ευρωβουλευτές θα αποφεληθούμε και θα προχωρήσουμε σε μια αποτελεσματική συνεργασία μέχρι την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, όποτε και αν είναι να συμβεί αυτό. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Ω προ το χρονοδιάγραμμα, υποβολή τροπολογιών ω τι 8 18 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΑΕΝΒΗ στις 20 ε, Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια στη δεύτερη του Νοεμβρίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καθαρή Ατμόσφαιρα για Όλους, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο ψηφίσματος βρίσκεται υπό διότι νομίζω τα περισσότερα μέλη αυτή τη επιτροπή, όταν ακούν για καθαρό αέρα, ε, πραγματικά ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερω, ειδικά όταν έχουμε με νομοθετικές πράξεις ε, που πρόκειται να εξεταστούν ή να περάσουν, γιατί δεν έχει τύχει σοβαρή διαχείριση στο θέμα αυτό και σε πολλά κράτη-μέλη τα πράγματα πάνε χειρότερα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το ψήφισμα. Νομίζω ότι καλύπτει όλους τους τομείς που θα έπρεπε να σχολιαστούν και θέλω απλώς να σταθώ σε μερικά σημεία. Να πω ότι στο πλαίσιο της δουλειάς που έκανα εγώ ως εισηγήτρια, για την ε, οδηγία που αφορούσε τα εθνικά μέτρα, ε, δείξαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορούμε να εργαστούμε σκληρά και να επιδιώξουμε και τους στόχους του Κοινοβουλίου μας. Η δυσκολία όμως που έχουμε σε μεγάλο βαθμό και χαίρομαι που βλέπω ότι το σχέδιο ψηφίσματος το καλύπτει αυτό και μάλιστα με καλό τρόπο, είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι αναγκαστικά η νομοθεσία, αλλά η υλοποίηση στα κράτη-μέλη και έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Σε κάποια κράτη-μέλη βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες και σε κάποια άλλη καμία απολύτως. Για τους πολίτες δεν υπάρχει καμία ε, πώς το αποζημίωση ε, για επιχειρήσεις και εταιρείε που ε, πρακτικέ του είναι σίγουρα επιζήμιε. Ακόμη και με τη βέλτιστη δυνατή ερμηνεία του τι συμβαίνει, ε, κανεί δεν έχει σταθεί ούτε καν στο γράμμα του νόμου. Αυτό είναι πλημέλημα των κρατών μελών ε, και μα ανησυχεί. Διότι μπορούμε να νομοθετούμε όσο μα αρέσει, αλλά τα κράτη-μέλη να μην εφαρμόζουν αυτά που νομοθετούμε. Ε, αυτό πρέπει να το δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω για την οδηγία για την καθαρή ατμόσφαιρα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα θα προκύψουν μάλλον στις αρχές της επόμενης χρονιάς και θέλω να είναι σαφές με το ψήφισμα αυτό. Ε, ελπίζω ότι κάποιοι από τους συναδέλφους θα θέλουν να γίνουν πιο στεναρό ακόμη το μήνυμα. Ελπίζουμε η οδηγία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας θα είναι πάρα πολύ εύρωστη και ότι θα ε, καθορίζει σημεία δράσης για το τι πρέπει να κάνουν στα επόμενα βήματα τα κράτη-μέλη. Ε, ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα παραμείνουν σοβαρά και δεν θα λένε το ένα πράγμα δημοσίω και μετά στην πράξη θα κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό κάνουν ω τώρα. Στην ατμόσφαιρα δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό. Όλοι έχουν δεσμευτεί τα 400.000 σε χρέος που υπάρχουν να τα αποπληρώσουν, αλλά υπάρχουν μια, ένα σωρό διαδικασίες παραβάσει και δικαστικές ε, ε, διαδικασίες οι οποίες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό το αναφέρει και το ψήφισμα. Και κάτι τελευταίο από πλευρά μου. Έχουμε εντοπίσει στο ψήφισμα συγκεκριμένα ζητήματα σε σχέση με τη γεωργία για το μεθάνιο και την αμμονία και η οδηγία ε, μιλά για την ατμόσφαιρα και πώς επηρεάζεται το όζον, αλλά και τις, ε, επιπτώσεις στην γη, την καλλιεργήσιμη γη. Δεν θέλουμε εδώ να ασκήσουμε πίεση στους γεωργούς, αλλά ανέκαθεν λέγαμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά εργαλεία για να τους βοηθήσουμε να κάνουν μια μετάβαση σωστή. Δεν είναι φτηνό εύκολο και θα πρέπει να καταβάλουμε σκληρότερες προσπάθειες για να μειωθεί η χρήση της αμμονίας, ας πούμε, στα, στην κτηνοτροφία. Προσπαθούν, δεν είναι ευθυνή εναλλακτική, αλλά θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Δεν είναι ένα θέμα που μας χωρίζει από τον κόσμο της γεωργίας. Πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας εδώ και να δουλέψουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Ντάνς τώρα από τους σοσιαλιστές. Λοιπόν, Βέβαια δεν σα εκπλήσει που και εμά ε, μας χαροποιεί το ψήφισμα αυτό, όπως λέει και η Τζούλη. Βεβαίω από καιρού καιρών πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης. Το ξέρουμε το θέμα, ξέρουμε την ε, διάσταση του θέματος. Κάθε χρόνο 400.000 ε, θάνατοι που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί και τρομερό κόστος για τα συστήματα υγείας λόγω της ε, κακής ποιότητας του αέρα. Και επειδή ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας υπήρξαν διάφορα νομοθετήματα, αλλά κάπως αποσπασματικά. Ορισμένα ε, είναι πιο φιλόδοξα, αλλά όχι. Και, όπως είπε και η Τζούλη, στην αρχή έχουμε πολύ καλές προθέσεις, ε, φιλόδοξες, αλλά κατόπιν υπάρχει μείωση. Μειώνονται οι φιλοδοξίες μας, είτε τα κράτη-μέλη, είτε άλλοι φορείς. Είναι υπεύθυνοι γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε κρίση. Η οποιαδήποτε επιτροπή, όποια και αν είναι η σύνθεσή της, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα αποσπασματικά βήματα ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή όλα μαζί θα λειτουργήσουν. Αυτό το ψήφισμα με σαφή αλλά σύντομο τρόπο μας λέει τι διαστάσεις έχει η πρόκληση που έχουμε ενώπιον μας. Φυσικά θα στηριχθεί από όλα τα κόμματα και ελπίζω να περάσει και το μήνυμα ότι και κάποιοι τομεί που πολιτικά είναι πιο ευαίσθητο ότι πρέπει να συμμετάσχουν να περάσει ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν. Προσπαθήσαμε και για, σε κάποια άλλα νομοθετήματα να επιβάλλουμε μέτρα στη Γεωργία που όμω ε, δεν έτυχαν ευρεία στήριξη όχι μόνο από του Γεωργού αλλά και από ορισμένα τμήματα εδώ τη επιτροπή μα. Κοιτάξτε, οι διαστάση του προβλήματο είναι πολύ σημαντικέ. Πρέπει να επιχειρήσουμε να μειώσουμε τι εκπομπέ ε, αμμονία και μεθανίου. Δεν καταλαβαίνουν ε, ορισμένοι πόσο συμβάλλουν οι γεωργικές εκπομπές, όχι μόνο στην Ήπεθρο αλλά και στις πόλεις, γιατί είναι πρόδρομοι ουσίες και μπορεί να παίξουν ρόλο στις ε, μισές περίπου επιπτώσεις ε, της μόλυνσης του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της γης μας είναι γεωργική. Πρέπει λοιπόν η χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής να σχετιστεί με το πρασίνισμα και κυρίως με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Υπάρχουν ήδη μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν. Δεν είναι φθηνά, αλλά έχουμε τους πόρους, έχουμε τη δυνατότητα παντού στην Ένωση να υπάρξει η επαρκής βελτίωση της κατάστασης. Αλλά δεν είναι εναλλακτική να μην κάνουμε τίποτα. Και οι μεταφορές βεβαίως πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα. Πρέπει να διορθώσουμε τις ε, επιπτώσεις του Dieselgate και θα πρέπει να είναι καθαρά τα οχήματα στους δρόμους μας οι μεταφορές είναι το πρώτο αίτιο της κακής ποιότητας του αέρα στις πόλεις. Και οι πόλεις έχουν τη δυνατότητα και τις εξουσίες να εισαγάγουν τα μέτρα που θεωρούν αναγκαία. Για παράδειγμα, περιοχές χαμηλών εκπομπών και άλλοι τρόποι περιορισμού πρόσβαση στα οχήματα. Παράλληλα, δηλαδή σε αντιστοιχεία με τις ανάγκες τους. Οι πόλεις ούτως ή άλλως λαμβάνουν πολλές πρωτοβουλίε. Εάν όλες αυτές αναχθούν σε ενωσιακό επίπεδο, θα συμβάλλουν ιδιαίτερα. Εάν λοιπόν ε, εξουσιοδοτήσουμε τις πόλεις για να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο, θα είναι θετικό. Κάτι άλλο για το πώ ε, αποδυναμώνουμε πολλές φορές ε, τα μέτρα μας. Από τότε που υπήρξε αυτή η οδηγία NECDR, 11 κράτη-μέλη, 11 κράτη-μέλη ζήτησαν προσαρμόσεις, ε, ε, ζήτησαν συγγνώμη, προσαρμογές στα ανώτατα όρια εκπομπών τους. Προς τα πάνω φυσικά. Οξύδια του αζότου κυρίως που εκπέμπονται από τα οχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε να υπάρξει μια τελική ημερομηνία για την κατάργηση του άνθρακα και επίσης του υδράργυρου που παίζει ε, τρομερά αρνητικό ρόλο για το νευρικό σύστημα, ιδιαίτερα και σε πολύ, ακόμη και σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Βεβαίω δεν είναι εύκολε αποφάσει αυτέ, αλλά η Επιτροπή πρέπει να τι λάβει. Και ελπίζω το κείμενο αυτό να ενισχυθεί περαιτέρω για να αποτελέσει βάση για μία πλήρη αλλά σύντομη οδηγία που θα προωθήσει κατόπιν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ επόμενη κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ. Σίγουρα όλοι γνωρίζουμε πόσο επιζήμιος είναι ο μολυσμένος αέρας, πόσο κακό μας κάνει η ατμοσφαιρική ρήπανση σε όλους τους πολίτες. Δεν χρειάζεται να μας πείσει κανένας γι' αυτό, είναι αυτονόητο. τώρα, θα ήθελα να επισημάνω ότι εσείς ε, ε, απευθύνεται έκκληση για αναβάθμιση των φιλοδοξιών και για όσο μεγαλύτερες, υψηλότερες δυνατές φιλοδοξίες, αλλά μέχρι τώρα πολλές χώρες δεν πληρούν καν τα κριτήρια και δεν ακολουθούν τους δείκτες που μέχρι τώρα έχουν προταθεί. Οπότε πώς θέλετε αν δεν τηρούμε τα μέχρι τώρα αποφασισμένα να ενισχύσουμε τις φιλοδοξίες. Άλλωστε το ελεκτικό συνέδριο στην ειδική έκθεση για το 2018 ε, που αφορά τις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την δημόσια υγεία λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπαση, φαίνεται από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ότι μέχρι τώρα δράσεις δεν έχουν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει λοιπόν αυτή η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου να αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη δράσης. Γιατί θα πρέπει πρώτα να τηρήσουμε τα μέχρι τώρα ε, μέτρα. Γιατί σίγουρα ε, τα αποτελέσματα της ατμοσφαιρικής ε, είναι και οικονομικά, χρειάζονται δαπάνες για τη δημόσια υγεία, αλλά και κοινωνικά, γιατί ε, δυσκολεύουμε τη ζωή των ε, συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας. Οπότε με βάση τα δεδομένα και τις αναλύσεις ε, να διαπιστώσουμε ότι η αυστηροποίηση των μέτρων δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν καν εφαρμοστεί τα μέχρι τώρα μέτρα. Αυτό θα πρέπει να μας γίνει μάθημα. Και η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι πολύ συχνά εμείς στην Επιτροπή Περιβάλλοντο μόνο μία λύση δίνουμε στα προβλήματα. Πιο φιλόδοξη στόχη. Στη συνέχεια όμως διαπιστώνουμε ότι παραβιάζονται ε, τα κριτήρια για, το, για την ατμοσφαιρική ρήπανση και αυτό το επιβεβαιώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που σημαίνει ότι μέχρι τώρα στόχοι είναι ανέφικτοι για πολλά κράτη-μέλη. Χρειάζονται λοιπόν μακροπρόθεσμες λύσεις, πολυσύνθετες, ε, που θα έχουν εξασφαλίσει όμως την απαραίτητη χρηματοδότηση. Αυτό πρότεινε η Πολωνία με την υλοποίηση ενός προγράμματος που είναι προτεραιότητα της πολωνικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα για τον καθαρό αέρα. Οπότε, ε, για το, την περίοδο 2014-2019 θα έχουμε περίπου 204 εκατομμύρια ευρώ και το συνολικό κόστος ε, της επένδυσης θα είναι πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. 2,4 συγγνώμη, εκατομμύρια και το συνολικό κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα με τις α, και την, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων ε, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο ανανεώσιμες πηγές καυσίμων με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες. Και χαίρομαι γιατί το ψήφισμα μιλάει για την συμβολή της τηλεθέρμασης και των δικτύων θέρμασης για την υλοποίηση των στόχων μας. Γιατί χάρη στην τηλεθέρμαση θα μειώσουμε αισθητά την ατμοσφαιρική ρήπανση. Γιατί τέτοια συστήματα τηλεθέρμασης ε, ε, αναγνωρίζονται σε λίγες χώρες, αυτές που έχουν τις πιο ακραίες καιρικέ συνθήκες και τους πιο ε, σκληρούς χειμώνες. Αλλά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης θα είναι πολύ πιο επιβαρυντικές, ιδιαίτερα στις πολυκατοικίες. Έτσι με την τηλεθέρμανση θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και την ποιότητα των καυσίμων και τις εκπομπές των αερίων στην ατμόσφαιρα. Θα πρέπει λοιπόν να εκτιμήσουμε το ρόλο της ε, τηλεθέρμανσης και στα πλαίσια της οδηγίας για τη μείωση εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρήπων και επίσης η ανάγκη δωρεάν αδειών. Το θέμα της τηλεθέρμανσης είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και ελπίζω εν καιρό να λάβουμε ορθολογικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Χάζενκα από την ΚΟΕ. En dat aantal zal alleen nog maar toenemen, want de huidige normen. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε ότι οι θάνατοι από την ατμοσφαιρική ρήπανση θα αυξηθούν. Γιατί στην Ευρώπη παρά είμαστε επίκης και δεν εφαρμόζονται αρκετά η νομοθεσία, δεν εφαρμόζονται αρκετά αυστηρά για να προστατευτούν οι πολίτες. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και μετά οχήματα και πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές από τον βιομηχανικό κλάδο, επιχειρήσης, επιχειρήσεις, ιδίως αστικές περιοχές. Η εντατική ε, κτηνοτροφία επίσης είναι μια σοβαρή πηγή ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Η κτηνοτροφία έχει σχέση και με την εκπομπή αμμονίας και μεθανίου, 40% της εκπομπής ε, αμμονίας και 94% του μεθανίου ε, οφείλονται στην εντατική κτηνοτροφία ακριβώς. Υπάρχει υψηλή συγκέντρωση των ουσιών αυτών και πολλές ασθένειες συνδέονται με την παρουσία τους στην ατμόσφαιρα. Πολλές επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η ε, εντατική κτηνοτροφία είναι και ένας από τους μεγαλύτερους λόγους, από τους σοβαρότερους λόγους, ε, ε, από τις πιο σοβαρότερες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, αλλά και αυτό των εκπομπών από τις μεταφορές. Θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα σοβαρό και να κάνουμε κάτι για τις εκπομπές. Δεν μπορούν να πνίγονται οι πολίτες μας από την κακή ατμόσφαιρα. Πρέπει να ενισχυθεί με κονδύλια η έρευνα και δεν γίνεται να κάνουμε ε, δώρα στην αυτοκινητοβιομηχανία με εξαιρέσει διαρκώ για τον τομέα αυτό. Πρέπει να υπάρχουν σαφείς και ξεκάθαρες αρχές ε, και κάποιες που να μας ε, κατευθύνουν. Θα πρέπει αυτοί που παίρνουν περισσότερο από του άλλου να πληρώσουν κάποια στιγμή. Και μεταξύ αυτών είναι και εντατική κτηνοτροφία. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. τελευταίο από την Ιευθυντή, η κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είμαι συνεισηγήτρια για το ψήφισμα αυτό, διότι ασχολείται με ένα θέμα ζωτικής σημασίας που απασχολεί τις πολιτικές μας προτεραιότητες, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Ιταλία. Οι πέντε αστέρες του Εγκοστέλη αυτή τη στιγμή έχουμε ως απόλυτη προτεραιότητα την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Γι' αυτό ε, έχουμε συμμετάσχει με πνεύμα συνεργασία στις προπαρασκευαστικές εργασίες που οδήγησαν στη σύνταξη του ψηφίσματος που σήμερα συζητάμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας και αυτό για μένα είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έχουμε από τις περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από αυτό, από την ε, του Πάδο, το Μιλάνο και τη Λομπαρδία από τι πιο ε, μολυσμένε περιοχέ στην Ευρώπη. Η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναπνέουμε έχει χειροπιαστά αποτελέσματα καθημερινά στη ζωή εκατομμυρίων πολιτών, στη Λομβαρδία και όχι μόνο. Πρέπει να υιοθετήσουμε ένα νέο παράδειγμα, ένα νέο πρότυπο ανάπτυξη. Διότι η πολιτική δεν μπορεί να αρνείται ακόμα το δικαίωμα σε, καθαρό, σε καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα στου πολίτε που το ζητούν επίμονα. Είδαμε οι περιοχές και οι κυβερνήσεις των περασμένων ετών να συνεχίζουν να εγκρίνουν ε, νομοθετικές πράξεις για τεράστιες διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, ε, υπερμεγέθη και να μην κάνουν τίποτα για την τιμωρία και την ε, αναχέτηση των ε, όσων ρηπαίνουν, κάτι που ήταν απαραίτητο. Η ποιότητα του ε, ατμοσφαιρικού αέρα λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί για να γίνουμε και αξιόπιστοι και σοβαροί. Δεν μπορούμε απλώς να λαμβάνουμε μέτρα όταν υπάρχουν κατεπίκουσε καταστάσεις, αλλά να δράσουμε σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, με τα κατάλληλα μέτρα και για να αντιμετωπίσουμε τις πηγές της ρήπανσης, όλους του τομείς τη οικονομίας και να αντιμετωπίσουμε τα οξύδια του αζότου και, όλες τις άλλες, ε, και όλους τους άλλους τύπους. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερχόμαστε αντιμέτωποι με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το, τις επιπαραβάσει διαδικασίες βάσει του άρθρου 10. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις δίκες για τις διαρκείς υπερβάσεις των ορίων στο διοξίδιο του αζότου και για να προφυλάξουμε τη ζωή των πολιτών, των περιβάλλων και τις μελλοντικέ γενιές όπως και αυτές που τώρα ζουν. Θα πρέπει να δούμε τι μέτρα να υιοθετήσουμε και τι επιλογές πρέπει να κάνουμε. Το συζητήσαμε και το συζητάμε και σήμερα και δεν υπάρχει σίγουρα μία κατεύθυνση. Είναι πολλοί οι τομεί που πρέπει να το ζητήσουμε να περάσουν σε μια μετάβαση και είναι αναπόφευκτο πλέον αυτό, όχι μόνο για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά για να επιδιώξουμε και του στόχου μα για τι κλιματικέ αλλαγέ. Το αναφέραμε ήδη. Οι μεταφορέ είναι ένας από τους τομείς που έχει συμβάλει στη διάρκεια του, ε, των ετών στην ένταση των ε, ατμοσφαιρικών ρήπων, διότι δεν έχει περιορίσει τις εκπομπές του με τη χρήση βρώμικων καυσίμων όπως το ντίζελ. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ε, δημόσιες συγκοινωνίες λοιπόν, εάν μπορούμε να δημιουργήσουμε ζώνες χαμηλών εκπομπών για τους πολίτες, εάν μπορούν να υπάρχουν περισσότερα οχήματα που να είναι καθαρά όπως ε, αυτά με τις μηδενικές εκπομπές το κατά πόσον μπορούμε να προωθήσουμε ε, καθαρότερες μεταφορές καθαρότερης ενέργειας. Πρέπει για όλα αυτά να βρούμε χώρο σε αυτό το ψήφισμα και θα ευχηθώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει παρόμοια διάθεση και σε μια άλλη μας ε, ε, απέτηση να έχουμε περισσότερο αυστηρά όρια για το PM2,5. Τα σωματίδια τα μικροσωματίδια 2,5 και τον περιορισμό τους. Ε, αυτό το έχουν ζητήσει επίμονα πολλές ενώσεις. Εδώ προκύπτουν σοβαρές ευθύνε και σίγουρα με την εντατική κτηνοτροφία και την εντατική γεωργία. Ελπίζω λοιπόν οι συνάδελφοι να ε, συνεχίσουν τη δράση για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης όχι μόνο στο, κέντρο των αστικών περιοχών αλλά και στις ε, περιαστικές περιοχές και στις περιφέρειες των πόλεων. Και όπως το αναφέραμε, είναι σημαντική η καταπολέμηση των σωματιδίων αλλά και του μεθανίου. Ε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που επιβαρύνει την ε, κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. And now I give the floor. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή, η κυρία Μανφρέντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρίε και κύριοι. Ε, καλωσορίζουμε αυτό το ψήφισμα το οποίο πραγματικά είναι ένα θέμα που για όλους μας είναι ιδιαίτερα καυτό, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο ε, διότι έρχεται να συζητηθεί σε μια στιγμή όπου πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Ε, ξέρουμε και την έκθεση του διακυβερνητικού πάνελ του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές και για την κατεπίγουσα ανάγκη να δράσουμε. Αυτό αφορά προφανώ το στόχο καθαρότερο ατμοσφαιρικό αέρα για όλου και αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών. Εδώ Πρέπει να πούμε ότι αυτό που συζητάτε είναι ότι ακόμη υπάρχει έλλειψη καλών αποτελεσμάτων, όπως είπατε οι περισσότεροι. Αλλά μην υποτιμάτε την προσπάθεια, την, ε, ε, το πόσα έχουμε ήδη πετύχει σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, όπου υιοθετήσαμε ε, μια πλήρη νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Χάρη στι κοινέ προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Εθνικών Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών, οι εκπομπές μειώθηκαν από 10 έως 70% ανάλογα με το, πώς, ε, με το τι συνέβαινε το 2000 και αυτό σε μια περίοδο οικονομικής αύξησης. Ε, παρόλα αυτά, είμαστε στο πλευρό σας και συμφωνούμε ότι ακόμη το φαινόμενο αυτό ε, οφείλει ευθύνεται για τον πρώιμο θάνατο εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και δεν πρέπει να υποτιμούμε το σημαντικό μας ρόλο ως ε, παγκόσμιων πρωταγωνιστών ε, στο θέμα αυτό. Όταν δούμε παγκοσμίως τη συμβαίνει με τη μετοσφαιρική ρήπανση, πραγματικά μας ανησυχεί να βλέπουμε ότι σε μερικά ευρωπαϊκά κράτη το επίπεδο του ατμοσφαιρικού αέρα είναι τόσο χαμηλή ποιότητα όσο σε κάποιε χώρε τη Αφρική, που είναι πραγματικά τραγικέ οι συνθήκε σε σχέση με το φαινόμενο αυτό. Πρέπει λοιπόν τα μέτρα μα να ενταθούν στην Ευρώπη διότι οι συνέπειε είναι σοβαρότητε σε πλανητικό επίπεδο. Μα ανησυχεί λοιπόν πολύ το τι συμβαίνει. Δεν ε, σημαίνει αυτό το ότι δεν έχουμε τέλεια αποτελέσματα, ότι δεν είμαστε και ε, οι πιο σοβαροί θεματοφύλακε των συνθήκων. 30 διαδικασίε επί παραβάση αναφέρατε στη ψήφισμά σα. Σε 20 κάτι πρέπει να. Εγώ πρέπει να διορθώσω τον αριθμό και να πω ότι είναι 20 αυτέ. Και η λογική μας για τη διαρκή αυτή ε, της επιβολής της νομοθεσίας είναι ότι ε, ο Επίτροπος Βέλα, ε, Βέλα λέει πάντοτε ότι ε, πρέπει να είμαστε αυστηροί στην επιβολή της νομοθεσίας με συγκεκριμένα δραστικά μέτρα. Ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να προβλέπει μέτρα για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, προκλήσεις. Και μόλις τώρα το συζητήσαμε για το πρόγραμμα LIFE, το LIFE που πρέπει να συνδυαστεί με άλλα εργαλεία του προπολογισμού. Ε, πολλά πρέπει να γίνουν για να υπάρξει αλλαγή. Να μην ε, αναφέρω τώρα τη γνωστή περίπτωση της περιοχής Μονοπόσκα, Πανοπόλσκα, Μαλοπόλσκα και να δούμε σε τι βαθμό μπορεί να ε, προχωρήσουμε και σε αυτό. Εδώ πρέπει να υπάρξει η σωστή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου όπου χρειάζεται, ιδίω για τι πηγέ τη ρήπανση. Ξέρετε πολύ καλά τι δουλειά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξαιτία του σκανδάλου Dieselgate προφανώς, κάτι που ε, θα, θα γινόταν κάποια στιγμή, γιατί κανεί δεν περίμενε ότι θα φτάναμε σε αυτά τα επίπεδα εξαπάτηση. Τώρα έχουμε τι απαιτήσει για τι δοκιμέ σε πραγματικέ συνθήκε οδήγηση και όλοι όσοι ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντο κοιτάζουν να έχουν πιο ειλικρινή διάλογο με όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχει πραγματική ανταλλαγή των βέλτιστων παραδειγμάτων και σύντομα θα διοργανώσουμε το δεύτερο φόρουμ για τον καθαρότερο αέρα και θα συνδυάσουμε την παρουσία των καλύτερων εμπειρογνωμόνων, αυτών που είναι πλέον επαείοντες στον τομέα αυτό, προσπαθώντας να προσφέρουμε χρηματοδοτική υποστήριξη στα κάτι μέλη που ζητούν οικονομική βοήθεια. Καλωσορίζουμε και το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στις εκπομπές από τον τομέα της γεωργίας και της κοινοτροφίας... και όπως και εσείς, τη γεωργία θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε σε ένα τομέα που πρέπει να οδηγηθεί προς την βιωσιμότητα. Ε, θέλουμε να δούμε πώς η Επιτροπή σας θα αξιολογήσει την πρόταση για την ΚΑΠ και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ζωτική σημασία στα μελλοντικά χρόνια. Αλλά αυτό με οδηγεί και σε μια άλλη παρατήρηση. Αντίθετα με ό,τι συνέβη στην περιοχή των ε, πλαστικών και τη σχετική ε, ε, τη κινητοποίηση, εδώ παγκοσμίω βλέπουμε να υπάρχει ε, κινητοποίηση. Στον τομέα του καθαρού αέρα δεν υπάρχει ανάλογη προβολή δεν υπάρχει ανάλογη ευαισθητοποίηση για τις πηγές του προβλήματος. Να εντοπίσουμε ξεχωριστά και μεμονωμένα την κάθε πηγή του προβλήματος και να δημιουργήσουμε την ανάλογη ενημέρωση και αντίδραση στο κοινό. Γι' αυτό πρέπει και το Κοινοβούλιο να συμβάλλει ώστε να ταρακουνήσουμε τον κόσμο με έναν τρόπο έτσι αρκετά έντονο ε, οι συσχετισμοί μεταξύ περιβάλλοντος και υγείας πρέπει να τονιστούν παντού. Και ε, αυτά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα συνεργαζόμαστε όλο ένα και στενότερα με τους συναδέλφους του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το ξέρετε, στις 30 Οκτωβρίου και μέχρι 1 Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη παγκόσμια σύνοδος για την ατμοσφαιρική ρήπανση και την υγεία θα είμαστε εκεί μαζί με πολλούς ε, επικεφαλείς και ηγέτες ε, του χώρου αυτού από όλο τον κόσμο και θα κοιτάξουμε την ενδυνάμωση, την ευθυγράμμιση, τη σχέση συνεργασίας, την, ε, τον συσχετισμό μεταξύ των ρηπογόνων πηγών και των συνέπειες στην υγεία. Θα πρέπει εδώ να συνδυάσουμε τη δράση μας σε όλους τους πολιτικούς τομείς. Είναι μια δική σας έκκληση αυτή, αλλά έρχεται η έκκληση τη στιγμή που το Σώμα των Επιτρόπων ε, συνάγει συμπεράσματα για το πώς μπορεί να βελτιώσει τη δομή διακυβέρνησης. Υπάρχει δυναμικό εδώ να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε το τι κάνουμε, εφόσον είμαστε ενωμένοι και βλέπω, θα πρέπει να ξέρετε ότι και τις εσωτερικές της διαδικασίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να τις εξορθολογήσει, αλλά θα πρέπει και στο Ευρωκοινοβούλιο να υπάρξει βελτίωση της εσωτερικής διάρθρωσης και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η θέση σε ισχύ των εθνικών οδηγιών για τα άνωτατα όρια είναι η πρώτη νομοθετική πράξη που ζητά από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν εθνικά προγράμματα για τον ατμοσφαιρικό αέρα ε, και να δουν τις πηγές ρήπανσης από όλους τους τομείς. Είναι μεγάλη αλλαγή στη διακυβέρνηση αυτό και πιστεύουμε ότι θα φέρει αλλαγή σε καθένα κράτος μέλος με τον ε, σκοπιμότερο τρόπο. Βεβαίως θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά πώς έχουν συνταχθεί τα εθνικά προγράμματα και θα σας ενημερώσουμε ως του χρόνου. Και πάλι τη, διαχείριση του θέματο αυτού μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Κάτι που κατά την ταπεινή μα άποψη είναι ένα θέμα που πάντοτε θα το διαχειρίζονται ε, επεύθυνοι πολιτικοί σε επίπεδο πρωθυπουργών τουλάχιστον γιατί αφορά όλε τι χώρε ταυτόχρονα. Καλωσορίζουμε το γεγονό ότι συνεχίζεται να τονίζεται τη σημασία τη μείωση ε, τη εκπομπή μεθανίου. Είναι πραγματική πρόκληση αυτό. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το 2014-2015 είχε προτείνει πρόταση για οδηγία με εθνικά ανώτατα όρια και προτείναμε να συμπεριληφθεί και το μεθάνιο. Ε, αλλά δυστυχώς ε, γίναμε μάρτυρες του γεγονότος ότι η συμφωνία ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ήταν αυτό το συγκεκριμένο αέριο να, να εξαιρεθεί από την ε, εν λογοδηγία. Κι όμως, βάσει της τότε δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μεθάνιο παρέμενε ε, μεταξύ των ουσιών που παρακολουθούμε. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το ε, Κοινό Ερευνητικό Κέντρο, με μια συγκεκριμένη μελέτη για τι επιπτώσει του μεθανίου στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το όζων και η μελέτη αυτή θα δημοσιευθεί σύντομα. Βάσει τη μελέτη αυτή και με τι προπορασκευαστικέ μα δράσει για την ετοιμασία τη τη για τη μακροπρόθεσμη ε, στρατηγική τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ε, θα κοιτάξουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα σχετικά πορίσματα και θα σα ενημερώσουμε για να δούμε πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Και πάλι λοιπόν, Πρόεδρε, ε, πολλέ ευχαριστίες για τη δουλειά σα. Είναι πραγματικά χρήσιμη και για μα και πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματικά περιθώριο για πολύ καλές ε, προσπάθειες συνεργασίας και για έγκαιρη δράση, διότι ξέρετε ότι ασχολούμαστε και για την, ε, ε, ασχολούμαστε και με την οδηγία για την ποιότητα του κυκλοφορώντος ατμοσφαιρικού αέρα. Θα σας ενημερώσουμε αναλόγως. Ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε θα ψηφίσουμε στην ΕΜΒΗ στις 26-27 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Τώρα το επόμενο θέμα. Προφορική ερώτηση. Για τους ε, επικονιαστές, η ενωσιακή πρωτοβουλία οι συνυπογράφοντες την προφορική ερώτηση. Ο κύριος λέει, από το ΕΛΚ πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα. Κοιτάξτε, εδώ και δεκαετίες ε, είμαι μελισσοκόμος. Ασχολούμαι λοιπόν με αυτό το θέμα. Την πρώτη η ιουνιου Επιτροπή πρότεινε επισήμω να ξεκινήσει δράση για να αντιμετωπιστεί η μείωση των επικονιαστών και ιδιαίτερα για του άγριου επικονιαστέ. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά την απαγόρευση τη ε, χρήση ε, σε ανοιχτό χώρο τριών νέων νοικοτινοειδών και αποδεικνύει τη δέσμευσή μα όταν θέλουμε για την προστασία των επικονιαστών που είναι πολύ διαφορετικά, διαφορετικοί επικονιαστές. και πρέπει να καταλάβουμε ότι τέσσερις στις πέντε σοδιές και άγρια λουλούδια εξαρτώνται από επικονιαστές για να ε, ε, αναπαραχθούν, καταλαβαίνουμε την ανάγκη δράσης. Όχι μόνο για την επιστηστική ασφάλεια και την παραγωγικότητα της γεωργίας, αλλά να διατηρήσουμε την βιοπικιλότητα. Η Επιτροπή προτείνει τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, βελτίωση της γνώσης ε, των λόγων για την μείωση των επικονιαστών. Δεύτερον, αντιμετώπιση των αιτίων αυτή της μείωση και τρίτον ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και συνεργασίες. Το Κοινοβούλιο έκανε λοιπόν ένα ψήφισμα, κάνει ένα ψήφισμα μάλλον και τονίζει την ανάγκη να μειωθούν περαιτέρω τα φυτοφάρμακα στους ε, βιότοπους των επικονιαστών και τα κράτη-μέλη και η Ένωση πρέπει να βοηθήσουν με μια ολιστική προσέγγιση όχι μόνο με προστατευόμενες περιοχές. Η βιοπικιλότητα χρειάζεται ευρύτερη προοπτική και όλοι οι επικονιαστές πρέπει να συμπεριληφθούν για να διατηρηθούν. Ο στόχο τη καλύτερη προστασία και η ε, δημιουργία νέων χαμηλού κινδύνου φυτοφαρμάκων και η απαγόρευση όλων των επικινδύνων φυτοφαρμάκων θα βοηθήσουν και οικονομικά και από πλευράς απασχόλησης. Καταλήγοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, την Τρίτη είχαμε μελισσοκόμους από την ε, Σλοβενία εδώ που έλαβαν φέτος ε, ένα ευρωπαϊκό βραβείο διότι ε, κήρυξαν τις 20 Μαΐου ως μέρα για την προστασία των μελισσών. Και είναι απόλυτα σαφές ότι η κατάσταση των μελισσών είναι πολύ καλός δείκτης για την υγεία του περιβάλλοντος. Το σχέδιο ψηφίσματος είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να στηριχθεί και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ που ήσασταν σύντομος. Οι άλλοι συνυπογράφοντες και αυτοί παρακαλώ να σεβαστούν τον χρόνο των τεσσάρων λεπτών. Οι περισσότεροι συνεισηγητές συν είναι παρόντε, οπότε θα έχουμε αρκετού ομιλητέ. η κυρία Κάντενμπαχ από πλευρά του ΕΛΚ Σωστά τα είπε ο Πέτερλε. Εγώ θα μιλήσω για τρία θέματα. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να δούμε το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Πρέπει να μας απασχολήσει και να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην βιοπικιλότητα. Γιατί μόνο έτσι θα διατηρηθούν και τα έντομα επικονιαστές μας. Που είναι πολύ σημαντικά και για την γεωργική μας παραγωγή και για γενικότερα για τα διάφορα είδη. διότι όλα τα έντομα αυτά κινδυνεύουν από την αύξηση της χρήσης των ε, φυτοφαρμάκων. Και στην ΠΕΣ το συζητήσαμε. Αλλά και εδώ υπάρχουν σημεία όπου μπορούμε να βοηθήσουμε στην επιβίωση των επικονιαστών εντόμων. Ευτυχώς στην Ευρώπη αυτά τα έντομα μας παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Ενώ σε άλλες περιοχές του κόσμου πρέπει να πληρώσει κανείς για τέτοια έντομα. Στη, στη Γαλιφόρνια για παράδειγμα μεταφέρουν με τεράστια φορτηγά μέλισσες δεξιά και αριστερά για να κάνουν ε, τον επικονιασμό. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε και στον κανονισμό για την προστασία των ειδών. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που έχουν ζητήσει τα κράτη για να χρησιμοποιούν νέο νοικοτινοειδή. Πρέπει να υπάρξει αυστηρότερη επίβλεψη. Γιατί λένε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις ανάγκης. Είναι όμως πολλές. Πολλά κράτη-μέλη. Δεν ιτολογούνται αυτές οι εξαιρέσεις που ζητάνε. Πρέπει να κάνει περισσότερα και η Επιτροπή και εμείς ως Κοινοβούλιο. Ελπίζω να υπάρξει ευρεία συνένεση για το ψήφισμά μας και καλό τους συναδέλφους να κάνουν συμπληρώσεις, τροπολογίες για να βελτιώσουμε ακόμη το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμές Μάκερ. Eh, eh, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους που συνέταξαν αυτό το εξαιρετικό ψήφισμα. Ξέρουμε όλοι ότι οι επικονιαστές ε, έχουν δύσκολη ζωή λόγω ε, διαφόρων παραγόντων. Ε, την κατάσταση της βιοπικιλότητας, τη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλες δυσμενείς συνθήκες. Δεν τονίζουμε όμως αρκετά τη σημασία των επικονιαστών και για την προστασία του περιβάλλοντο αλλά και για την οικονομία μα. Το 2016, στην έκθεση μα για την επικοινότητα, είχαμε απευθύνει συγκεκριμένη έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για του επικονίαστε. Και ε, το ψήφισμα που έχουμε επιτάπητος έχει πολλά θετικά στοιχεία τα οποία τα καλωσορίζουμε. Όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Η πρωτοβουλία απαιτεί να δοθεί συγκεκριμένη προσοχή στις ε, ειδικέ ε, τις ειδικές ε, συνθήκες και αίτια της εξάλληψης των επικονιαστών. Θα πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του και το ψήφισμα να συνεχίσει να αναφέρει σωστά τις πηγές του προβλήματος, όπως ε, την χρήση φυτοφαρμάκων που έχει να κάνει με την ΚΑΠ. Ευχαριστώ, κυρία Ρίση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό είναι πραγματικά κρίσιμο, το είπαν και οι προλαλήσαντες και ο κύριος Δεμεσμάκερ μας υπενθύμησε ότι ήδη ζητούσαμε σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2016, ζητούσαμε δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι τεράστιο το διακύβευμα. Δεν θα επαναλάβω τα νούμερα, τα γνωρίζουμε όλοι. Ένα άρθρο που αφορά το Βέλγιο, την πατρίδα μου, και αναφέρεται θνησιμότητα μελισσών από τον περασμένο ε, χειμώνα άνευ προηγουμένου επίπεδα θνησιμότητας ε, μελισσών στο Βέλγιο. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ε, η πρωτοβουλία του Ιουνίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίζει καλύτερη γνώση του φαινομένου. Καλή διάγνωση, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, να δούμε τα αίτια του προβλήματος, που έχουμε κάπως εντοπίσει. Χθε διάβασα στο γραφείο μου μία μελέτη ε, στο, από τη Σουηδία στο περιοδικό Biological Conservation. Εκεί αναφέρεται ότι η σταθερότητα των πληθυσμών επικονιαστών είναι συνάρτηση της ε, έντασης ε, της γεωργίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε πού είναι τα μέτρα που αντιμετωπίζουν τα αίτια της μείωσης των μελισσών, αλλαγή χρήσης γης στην Ευρώπη, εντατικές μορφές γεωργίας, χρήση φυτοφαρμάκων. Αφιερώσαμε στην Επιτροπή μας ένα ολόκληρο απόγευμα στην επιρροή των φυτοφαρμάκων ε, στις μέλισσες. Θα πρέπει να στραφούμε προς μη χημικές μεθόδους ή σε φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου και να καταργήσουμε τα νεονικοτινοειδή. Επίσης, ε, τον περασμένο Ιούνιο είχαμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μελισσών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχει δυνατότητα συνεργασία με και γεωργών. Υπάρχουν εταιρικέ σχέσει ε, αμοιβαίω επωφελεί για τους ενδιαφερόμενους και για τα οικοσυστήματά μας. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αίτια του προβλήματος, να ενθαρρύνουμε τις απαραίτητες δράσεις και αυτό ζητούμε και στο ψήφισμά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ρης. Από την ΚΟΕ τώρα, η κυρία Κόνετσνα. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι ε, πελαγοδρομούμε. Είχαμε πολλές ε, μελέτες για τη μείωση των επικονιαστών ε, και γνωρίζουμε το φαινόμενο, αλλά τι κάνουμε με τα πορίσματα των μελετών, τα εφαρμόζουμε και τις συστάσεις. Γιατί τα εντομοκτώνα, τα φυτοφάρμακα είναι αποδεδειγμένος επιζήμια για την υγεία των μελισσών. Κι όμως βλέπουμε ότι πολλά έχουν εγκριθεί για την επόμενη περίοδο. Ε, και μάλιστα συστηματικά εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας για τις εγκρίσεις ε, νέων φυτοφαρμάκων. Κάθε φορά στην Επιτροπή μας ε, το τονίζουμε. Τι κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνει τη μείωση των επικονιαστών, αλλά μένει με τα χέρια σταυρωμένα. Θα πρέπει να απαγορεύσουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων. Είναι η μόνη λύση για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο οι μέλισσες αντιμετωπίζουν νόσους, ιούς, ε, ε, ρήπανση από αλουμίνιο, φυτοφάρμακα. Κάθε χρόνο διαπιστώνουμε τα προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, ούτε να, να τα αντιμετωπίσουμε. Οπότε κρατάμε τα πράγματα ως έχουν, δεν βλέπουμε καμία αλλαγή και απλώς γινόμαστε ανήμποροι μάρτυρες της μείωσης του πληθυσμού των μελισσών. Γνωρίζουμε ότι τα φυτοφάρμακα με νεονεκοτενοειδή έχουν επιζήμια αποτελέσματα για το περιβάλλον και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε στα χωράφια μας. Πολλές χώρες δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν εξαιρέσει παρόλο που ισχύει η πανευρωπαϊκή απαγόρευση των νέων νοικοτινοειδών. Και μάλιστα σε... ούτε καν η απαγόρευση θα ήταν η λύση η πλήρης απαγόρευση των νοικοτινοειδών. Σε λίγο το μέλι θα γίνει είδος πολυτελείας. Και θα έχουμε και κρίση στην παραγωγή τροφίμων, γιατί δεν θα γίνεται επικονίαση των φυτών και άρα δεν θα έχουμε καλλιέργεια. Ελπίζω να εγκριθεί το ψήφισμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην περιοριστεί σε κενές υποσχέσεις ε, στις ε, προφορικές μας ερωτήσεις, αλλά θα αναλάβει επιτέλους δράση. Το πρόβλημα που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η αοριστία που χαρακτηρίζει τους στόχους της. Θέλουμε σαφείς στόχους και κα... κατηγορηματικές απαγορεύσεις και επίσης εφαρμογή των απαγορεύσεων από τα κράτη-μέλη. Θέλουμε τη βοήθεια των κρατών μελών που θα πρέπει να αποφύγουν την προσφυγή στις εξαιρέσεις. Θέλουμε πραγματικά να επέλθει μια τραγωδία μία καταστροφή πριν αναλάβουμε δράση. Και δεν έχουμε μόνο τη μείωση των επικοινωνιαστών εδώ, έχουμε και άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντορνανό. Ντορνανό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήμουν η συγγήτρια της γνωμοδότησης της ΕΒΗ για το μέλλον του της μελισσοκομίας πριν από ένα χρόνο και διαπιστώνω ότι το σχέδιο αυτοψηφίσματος που αφορά τους ο γενικό ε, ακολουθεί μια σωστή άγουσα. κάνει μια διαυγή διάγνωση του πολυσύθητου προβλήματος των εντόμων επικονίας στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξη και θέλω να είμαι επικοδομητική, αλλά ο αγώνας για να σώσουμε τα έντομα επικονίασης ε, δεν έχει κερδιθεί ακόμη. Τώρα, για τα νεονικοτινοειδή. Έχουμε τις τρεις ουσίες που αναφέρονται στο ψήφισμα, που θα πρέπει οπωσδήποτε να απαγορευτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019. Και παρόλα αυτά, παρά την ολοσχερή απαγόρευση, θα επιτρέπεται κατά εξαίρεση χρησιμοποίησή τους στα θερμοκήπια. Υπάρχει πρόβλημα όμως με την ρήπανση των εδαφών και των ετροφόρων ε, οριζόντων, γιατί χρησιμοποιούνται παρόλα αυτά για την άρδευση. Ε, το Βέλγιο μάλιστα δήλωσε ότι θα εξετάσει την πιθανότητα χορήγηση απαλλαγής και θα καταθέσει έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην είμαστε αφέλεις. Πολύ πιθανό και άλλες χώρες μέλη να ζητήσουν εξαιρέσεις. Κάτι που θα εκμηδενήσει τα αποτελέσματα αυτής της απαγόρευσης των νεονικοτινοειδών που ήδη είναι περιορισμένη εμβέλειας. Σε ό,τι αφορά τα άλλα νεονικοτινοειδή, Αυτά τα τρία δεν αναφέρονται δυστυχώς από την ε, ευρωπαϊκή απαγόρευση. Το ίδιο και για τη και φίλοι προ τη Επίσης είναι ε, εξίσου επιβλαβής ουσίες με τα νέα νοικοτινοειδή. Όπως λέω σε μια τροπολογία μου πριν από ένα χρόνο, η γλυφοσάτη επίσης ε, αποδείχθηκε ότι είναι τοξική για τις μέλισσες. Δεν επιτέλους ώρα να την καταργήσουμε παρά τους υπερμάχους που έχει αυτή η ουσία. Εν πάση περιπτώσει, το, το ψήφισμα είναι θετικό. Θα καταθέσω όμως και άλλες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ε, υπόλοιπους συντάκτες του ψηφίσματος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκοντίνα. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Να μην επανέλθω στην κακή κατάσταση των επικονιαστών στην Ευρώπη. Το ψήφισμά μας είναι σαφές. Μειώνονται. Αλλά πρέπει να δούμε τι ποσοστό. 40% από τα ίδια επικονιαστές είναι, ε, απειλούνται με εξαφάνιση και 40% της γεωργικής μας παραγωγής ε, κινδυνεύει εάν εξαφανιστούν και κινδυνεύει η επιστησική μας ασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν αντιφάσεις μεταξύ των ε, αναγκών του περιβάλλοντος και της γεωργίας. Πρέπει να διατηρήσουμε τους πληθυσμούς των επικονιαστών. Αλλά υπάρχει και ένα μεθοδολογικό θέμα. Όταν ε, θα συμφωνήσουμε σε ένα φιλόδοξο κείμενο για να διατηρήσουμε αυτό το ζωτικό δεσμό μεταξύ επικονιαστών και βιοπικιλότητας για την υπεθρό μας και για τη γεωργία μας, θα ε, πούμε τα ίδια, τα ίδια παράνο, παράλογα που κάναμε παρά τις αντιρρήσεις που είχα εγώ. <coughs> Υπάρχουν τα νεονικοτριδοειδή νέας γενέας που στη Γαλλία έχει απαγορευτεί. Ενώ η Επιτροπή μας δεν είχε το θάρρος να το απαγορεύσει το 2015. Υπάρχει και το ασεταναμιπρίντ που βρίσκουμε κατάλοιπά του στα γεωργικά προϊόντα. Αλλά δεν υπάρχει πλειοψηφία εδώ μέσα για να προστατεύσουμε στην πράξη του επικονιαστές. Επίση, <clears throat> υπάρχει μια πρόταση στο 11 του ψηφίσματο μα την οποία στηρίζω, να απαγορευτεί πλήρω κάθε μορφή νέων νοικοτινοειδούς. Αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς, συνάδελφοι. Πρέπει να απορρίψουμε τις μελλοντικέ προτάσεις της Κομισιόν που δεν συμφωνούν με αυτήν την κατεύθυνση. Πέρα από πολιτικές διαφορές, Πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε τους επικονιαστές. Και θα κάνω τροπολογίες, ούτως ώστε οι ε, ενώσεις οι οποίες θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τα νέα νοικοτινοειδή να απογορευτούν και αυτές. Ευχαριστώ, Επιτροπή. Η κυρία, ο κύριος Ντελγκάντου Ρόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που καταλαβαίνουν όλοι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μείωση των επικονιαστών. Που δεν είναι θέμα μόνο μείωση των επικονιαστών, είναι θέμα μείωση τη βιοπικιλότητα. Ε, κινδυνεύουν διάφορα έντομα. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να αποφελούμεθα από τι υπηρεσίε των ε, πολυπλόκων οικοσυστημάτων. Του επικονιαστέ του καταλαβαίνει όλου το ρόλο τους και τα ωφέλη τους για τη γεωργία. Τώρα να τα δούμε σε ένα πλαίσιο. Η Ενωσιακή Πρωτοβουλία για τους Επικονιαστές εστιάζει στους άγριους επικονιαστές. Δεν ασχολείται με όλους τους επικονιαστές. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ουσιώδεις ανάγκες. Αλλά η πρωτοβουλία αυτή συμπληρώνει υπάρχουσα μέτρα για τη γεωργία, για την υγεία των μελισσών. Και θέλει να συμμετάσχουν και οι μελισσοκόμοι στην προστασία και των αγρίων επικονιαστών. Βεβαίως εστιάζουμε στην γνώση, γιατί υπάρχουν κενά στη γνώση μας, αλλά το επίπεδο γνώσης που ήδη έχουμε σημαίνει μας επιτάσσει συγκεκριμένες δράσεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη μείωση των επικονιαστών. Η πρωτοβουλία εστιάζει στους βασικούς, όπου χρειάζονται επιπλέον προσπάθειές μας, που να επιφέρουν προς τη θεμένη αξία. Για παράδειγμα, να ενισχύσουμε τα προβλήματα με την μείωση του χώρου ε, των οικοτόπων αυτών των αγρίων επικονιαστών. Αλλά υπάρχουν βέβαια και άλλοι κίνδυνοι. Ένας για παράδειγμα είναι η κλιματική αλλαγή. Αλλά οι απόψεις των ειδικών που ρωτήσαμε δεν μας έκαναν συγκεκριμένες προτάσεις για την περίπτωση των επικονιαστών. Είναι ένα σφαιρικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν πρόκειται να τροποποιήσει την, την πολιτική μας για την κλιματική αλλαγή. Δεν θα επέφερε βελτίωση για τους επικονιαστές. Οι ασθένειες, για παράδειγμα, από ό,τι ξέρουμε, κυρίως αφορούν τους ελεγχόμενους επικονιαστές δεν έχουμε πληροφορίες για την επίπτωσή τους στους άγρους επικονιαστές. Ε, το ίδιο ισχύει και για βαρέα μέταλλα, την ε, μόλις από το φωτισμό, την ατμοσφαιρική ε, ρήπανση. Δεν γνωρίζουμε πώς επηρεάζουν τους άγρους επικονιαστές, αλλά δεν μπορούμε να λάβουμε μέτρα. Είναι η πρώτη συνολική δράση της Ένωσης για τους άγρους επικονιαστές. Θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν κάποιες θεμελιώδεις διαδικασίες. Πρέπει να υπάρχει συστηματική παρακολούθηση των άγριων επικονιαστών για να δούμε την κατάσταση και τις τάσεις. Δεν ξέρουμε το ρυθμό μείωσης τους. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε λοιπόν την επίπτωση των δράσεων που θα αναλάβουμε, δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρξει ένα σύστημα κοινών προδιαγραφών για την αξιολόγηση της επίπτωσης των ε, μέτρων μας επί των αγρίων επικονιαστών συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων γεωρικής πολιτικής, επί της οποίας γεωρικής πολιτικής προσθέτω. Στην ε, πρότασή μας για την ε, ΚΑΠΑΓΑΜΑΠΗ μετά το 2020 κάνουμε και πολύ καλές προτάσεις. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο είπαμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η επίτευξη μέσω της γεωρικής πολιτικής των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης. Να προστατεύσουμε περισσότερο τα οικοσυστήματα, τους βιοτόπους, την Ήπεθρο, τα τοπία. Και αυτή η νέα ΚΓΠ που θα περάσει από τη συμμόρφωση προς την επίδοση θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τι προτάσει του που να καλύπτουν και το ενδεχόμενο μόλι από τον ένα τομέα στην άλλη. Θα υπάρχουν βεβαίω κάποια οικοσυστήματα που θα είναι θελούσια για του γεωργού υπό τον πρώτο πυλώνα, αλλά μπορεί να έχουμε και οικοπρογράμματα για του επικονιαστέ. Και βεβαίω σε συνεργασία και με την ε, ε, νομοθεσία μα για το περιβάλλον. Όλα αυτά θα συνδυαστούν. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τι φιλόδοξα περιβαλλοντικέ προτάσει τη Επιτροπής, γιατί αυτό θα ωφελήσει και τον τομέα που συζητάμε εδώ. Και γενικότερα την ε, βιοπικιλότητα. Για τα φυτοφάρμακα. Βέβαια, δεν θα υπάρξει σημαντική ε, μεταρρύθμιση μέσω αυτής της πρωτοβουλίας της ε, πολιτικής μας για τα φυτοφάρμακα. Αλλά Επανέρχομαι στις ε, προτάσεις για την γεωργική πολιτική. Θέλουμε να υπάρχει βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων. Είναι στόχος. Υπάρχουν και δείκτε για την πολιτική μας για τα φυτοφάρμακα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να βελτιώσουν τα εθνικά προγράμματα δράσης για να εφαρμοστεί η οδηγία για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων. Υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτε για τη μείωση των κινδύνων, Εμεί ω Επιτροπή θέλουμε να μειωθούν οι κίνδυνοι από τα φυτοφάρμακα. Και όχι να πούμε γενικά να μειωθεί ο όγκος χρήση φυτοφαρμάκων. Απλώς. Θέλουμε να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέσω μείωση της χρήση των φυτοφαρμάκων. Θέλουμε, για παράδειγμα, να υπάρξουν συγκεκριμένοι δείκτες κινδύνου που συζητάμε τώρα με τα κράτη-μέλη για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε και σε κρατικό και σε ενωσιακό μέλλον για να δούμε και μετά στο μέλλον τι πολιτικές θα προτείνουμε. Για να υπάρχει σωστή εφαρμογή της οδηγίας αυτής πρέπει να έχουμε μη χημικές μεθόδους ελέγχου των παρασίτων. Αυτό θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους χρήστες των φαρμάκων και είναι μάλλον από τον Ιανουάριο του 2014. Και στις εκθέσεις που έχουμε κάνει επικρίνουμε τα κράτη-μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει τις αρχές της ολοκληρωμένης πολιτικής ελέγχου των παρασίτων. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να διορθώσουν αυτές τις ελλείψεις. Να έχουμε καλύτερη εφαρμογή λοιπόν των ε, μη χημικών μεθόδου, μεθόδων ελέγχου των παρασίτων. Για τις μέλισσες έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο για να τις προστατεύουμε από τα φυτοφάρμακα, περιορισμοί της χρήσης τριών νέων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε θερμοκήπια. Αλλά πρέπει να θεωρήσουμε βεβαίως ε, ρωμαλαία αυτές τις ε, οδηγίες για να, υπάρξουν, για να υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις. Δεν λέμε Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται περαιτέρω νομοθεσία για τις μέλισσε. Επίσης, ε, εμείς δεσμευόμεθα για την ενέργεια 7β του προγράμματος. Να υπάρξει ένα σχέδιο εφαρμογή <clears throat> για το έγγραφο καθευτηρίου γραμμών της ΕΦΣΑ για τα προϊόντα που εισάγονται και τι επιπτώσει έχουν στις μέλισσε. Είναι προτάσει που τι συζητάμε τώρα με τα κράτη-μέλη. Άρα Βέβαια δεν μπορεί να περιμένουμε μέσω της πολιτικής επικονίας το να αλλάξουμε όλες τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, αλλά προσπαθούμε να ενισχύσουμε την προστασία των επικονιαστών και ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και ευρύτερα προβλήματα. Μείωση της βιοπικιλότητας στις γεωργικές γέες και γενικότερα το πρόβλημα της ε, επιδείνωσης της κατάστασης των ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να δούμε και το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 15 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΒΙ στις 26 και 27 Νοεμβρίου ή στις 26 ή στις 27. Η ψηφοφορία στην Ολομέλη θα γίνει το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση και να πάμε στο επόμενο θέμα που είναι και πάλι προφορική ερώτηση που συνοδεύεται από ψήφισμα με τίτλο ενδυνάμωση της ψηφιακής μετάβασης, της υγείας και της οικονομικής περιθαλψής στην ενιαία ψηφιακή αγορά και δίνοντας ε, τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στην ψηφιακή κοινωνία. Να ξεκινήσω δίνοντας το, λόγο στους ε, συντάκτες της ε, ερώτησης και του ψηφίσματος. Πρώτα απ' όλα για το έλκο ο κ. Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Ρόζα που είναι και παλιός ε, συνάδελφος. Ε, Πιστεύουμε ότι τα ψηφιακά μέσα είναι ένας τρόπος να πετύχουμε ευημερία, καλή υγεία και ε, ποιότητα ζωή διαβίωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ασχοληθήκαμε με διάσκεψη, σε διά, διάσκεψη ε, ημέρες για τα μεγάλα δεδομένα το δυναμικό των ε, big data για να βελτιώσουν τον τομέα της υγείας είναι πολύ μεγάλο για να στηρίξουμε τις δημόσιες πολιτικές υγείας, να έχουμε ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη και να μειώσουμε το κόστος για την υγεία. Οι ευκαιρίες της ψηφιοποίησης είναι τεράστιες. Η ιατρική πρακτική επιτρέπει να υπάρχει διεθνή συνεργασία για την αναχέτηση των ασθενειών και ε, κατάλληλη αγωγή που να διαδίδεται εκεί που πρέπει για να αντιμετωπιστούν οι επιδημίες. Επίσης, προκλήσεις υπάρχουν στον χώρο των ψηφιακών λόγω της προσωπικής, της απόρριτης φύσης των πληροφοριών που ε, έχουν να κάνουν με το ιστορικό των ασθενών, πρέπει να είναι μυστικό. Ε, προσπαθούμε με τον κανονισμό προστασίας των δεδομένων να φροντίσουμε και τον ιδιωτικό βίο των ασθενών, ενώ τα χρήσιμα δεδομένα θα πρέπει να ανταλλάσσονται για σκοπού έρευνα και προστασία. Νομίζω το μέλλον θα μα πει σε τι βαθμό πετύχαμε το σωστό σημείο ισορροπία. Επιπλέον, σε σχέση με τις προκλήσεις τη της προστασίας των δεδομένων των ασθενών, έχουμε και άλλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, όπως τις υποδομές για τα δεδομένα, διότι οι βάσεις δεδομένων για την υγεία είναι πολύ κατακαιρματισμένες και δεν είναι ενοποιημένες. Ταυτόχρονα, οι ευκαιρίες για τη χρήση των μεγάλων δεδομένων απαιτούν ε, νομικά και πολιτικά μέτρα στον τομέα της ψηφιακής υγείας και της ε, φροντίδας σε σχέση με τα δικαιώματα των ασθενών και κυρίως για την ανταλλαγή των δεδομένων, την πρόσβαση σε αυτά και την διευκόλυνση της υγείας των ασθενών και την ε, δουλειά των ε, υπευθύνων στον τομέα υγείας. Ηλεκτρονική υγεία. Προκλήσεις και δυσκολίες αλλά και ευκαιρίες παρόλα αυτά υπάρχουν και ευκαιρίε. Η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να συμμετέχουν όλοι, να συμμετέχουν όλοι και να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ασθενών. Θα πρέπει όχι μόνο οι εταιρείε οι τεχνολογικές εταιρείε να εξυπηρετούνται, ε, το ίδιο και οι νεότεροι ασθενεί και οι υπεύθυνοι στο χώρο υγείας, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν τόσο καλά τα ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να διατίθενται σε όλου και να υπάρξει αλλαγή στο πρότυπο που χρησιμοποιούμε. Το σχέδιο ψηφίσματο που παρουσιάζουμε σήμερα επιτρέπει την ηλεκτρονική μετάβαση στο τομέα τη υγεία και τη οικονομική περιθαλψή στην ενιαία αγορά, δίνοντα δυνατότητα στου πολίτε και επιτρέποντα να ε, χτίσουμε το μέλλον. Καταγράφει την σωστή πρόσβαση και την ε, ε, ανταλλαγή των πληροφοριών για την υγεία την, ε, ε, τον συνδυασμό των δεδομένων για την καλύτερη ε, εξυπηρέτηση των ασθενών και την ενδυνάμωση των υπευθύνων για την υγεία στην διαχείριση των δεδομένων αυτών, στον τομέα τη πρόληψη και τη πληροφόρηση για την υγεία, λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Στου καιρού των ψευδών ειδήσεων του λαϊκισμού και τη κινδυνολογία, όπως είδαμε πρόσφατα και με τα εμβόλια, η προσπάθεια για τέτοια σωστή πληροφόρηση είναι ύψης της σημασίας, πιστεύω. Επίσης πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αρχές θέλουν να βοηθήσουν και όχι να δημιουργήσουν περισσότερα εμπόδια. Αυτό θα τους καταστεί σαφές εάν η ηλεκτρονική υγεία χρησιμοποιείται για να καλύπτουμε τα κενά της διαρκούς και ομαλής ε, προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών όπως χρειάζονται οι πολίτες. Τέλος, να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές μου για την εξαιρετική μας συνεργασία Θα περιμένω λοιπόν ε, τις ε, συνεισφορές σας για να βελτιώσουμε το σχέδιο του ψηφίσματος και η επόμενη φάση είναι η υποβολή τροπολογιών. Θα ανακοινώσει ο πρόεδρος την προθεσμία φαντάζομαι μετά. Ευχαριστώ πολύ και μετά, και μετά για τους σοσιαλιστές ο κύριος Ζωρίνιου. Παρακαλώ και εσείς να μείνετε στα τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το ψήφισμα που συζητούμε ορίζει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες του Ευρωκοινοβουλίου για ένα θέμα που είναι κεντρική σημασία για την κοινωνία μας. Η ψηφιακή μετάβαση και ο αντίκτυπος στην εξέλιξη του τομέα της υγείας. Τα συστήματα υγείας πρέπει να επικεντρωθούν στο να ε, καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών, των ασθενών. Οι νέες τεχνολογικές λύσεις και τα νέα μέσα πρέπει να ενισχύσουν αυτήν την αρχή, αυτή την επιδίωξη τα συστήματα υγείας που επικεντρώνονται στις ανάγκες των ασθενών πρέπει να εξερευνούν τις ευκαιρίες και να φροντίζουν για την ενεργό συμμετοχή όλων. Θα πρέπει να υπάρξουν δίκτυα συμμετοχής, κατά τρόπο ώστε οι χρήστες να ε, μπορέσουν να εξοπλίσουν τα μέσα και να υπάρχει ε, μια καθολική και ανεπίσημη συμμετοχή. Θα πρέπει τα συστήματα να είναι διαλειτουργικά εύχριστα και ε, λειτουργικά. Οι πληροφορίες να συγκεντρώνονται σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο από τι αρχέ και να προφυλάσσονται όπω πρέπει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από τη δική μου τη σκοπιά. Μια άλλη προτεραιότητα είναι να τα δεδομένα με τρόπο ασφαλή σε διασυνοριακό επίπεδο. Διότι περισσότερα δεδομένα θα επιτρέπουν να βρίσκονται καλύτερε αποκρίσει για περισσότερου ανθρώπου, περισσότερου πολίτε. Η, μετάβαση, η σταδιακή μετάβαση στην ψηφιοποίηση πολλών συστημάτων υγεία έχει να κάνει και με το πόσο θα είναι αποτελεσματικέ εταιρικέ σχέσει μεταξύ των διαφορών εμπλεκομένων στο όλο σύστημα, τι δημόσιε αρχέ και του ιδιωτικού φορεί. Ο δρόμο για να βρούμε καθόλου καθολική πρόσβαση στην ψηφιοποίηση της υγείας για όλους τους πολίτες θα είναι ένα κίνητρο ώστε η Ευρώπη να ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ώστε όλοι να αποκτήσουν ψηφιακές δυνατότητες. λόγω χάρη να ορίσουμε σωστά τους όρους και τις τις ιδιότητες που χρειάζονται για να μπορεί κανείς να υποφεληθεί και να έχει πρόσβαση θα πρέπει να προωθήσουμε την υγεία, διότι θα πρέπει ε, να ενταχθεί σωστά στον, ε, στην ενιαία ψηφιακή αγορά και να μην τα αφήσουμε αυτό στην ελεύθερη βούληση των αγορών. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες προς όφελος των πολιτών και να προσφερθούν υπηρεσίες ε, με κάποιο νόημα, ώστε να καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Η δουλειά που κάναμε εδώ με τους συνσυντάκτες ε, οδήγησε σε ένα ψήφισμα που πιστεύουμε ότι προσφέρει την θετική, μια θετική συμβολή στον δρόμο που μόλις σας ανέφερα. Next is Ms. Krupa. Ευχαριστώ κυρία Κρούπα. Ευχαριστώ. Αυτό το σχέδιο ψηφίσματος θέτει κάποιες ερωτήσεις, επισημαίνει κάποιες προκλήσεις. Καταρχήν, ποιοι είναι οι άμεση ε, δικαιούχοι αυτού του εγγράφου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ε, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στις διάφορες χώρες ε, και αυτό θα δηλαδή θέλω να το διορθώσω με τροπολογίες, ώστε οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ε, είναι επιφορτισμένες με την διόρθωση του συστήματος και την προστασία των πολιτών που είναι δικαιούχοι αυτού του συστήματος. Και η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Και θα πρέπει να κάνουμε ένα σαφή προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων ε, και των ανεξάρτητων ε, φορέων που θα είναι υπεύθυνε για τη διατήρηση και για την επεξεργασία των δεδομένων. Για όλα αυτά τα θέματα θα καταθέσω τροπολογίες και σίγουρα το δικαίωμα των ασθενών υπερτερεί του δικαιώματος της ε, χρήσης των δεδομένων. Επίσης, ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μερικές φορές ε, θα έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ των ασφαλιστικών ε, εταιριών και των ε, ιατρικών Ινστιτούτων. Παρόλο που το ψήφισμα στα σημεία 3 7 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων. παρόλα αυτά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα διεκδικούν όλο και περισσότερα στοιχεία και εκεί δημιουργείται πρόσφορο έδαφος ε, για απειλές. Το θέμα είναι ποιο όργανο, ποιος φορέας θα είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Θα πρέπει ε, να έχουμε χέγγια στο μέλλον ότι δεν θα δημιουργηθεί μια κεντρική βάση ε, για, την, ε, για τα δεδομένα των ε, πολιτών και την κατάσταση υγεία τους, υγείας τους. Επίσης, τι Ινστιτούτα θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα. Για παράδειγμα, φαρμακοβιομηχανίες θα έχουν τέτοια πρόσβαση. Ή τα Υπουργεία Υγείας, οι, οι ασφαλιστικές εταιρείε. Σε ό,τι αφορά τις φαρμακοβιομηχανίες, αυτό είναι μια άλλη πρόκληση και, απειλή που ίσως δημιουργείται. Γιατί ε, σε πολλές χώρες ε, επιστρέφονται τα φαρμακευτικά έξοδα, είτε μερικά είτε πλήρως, αλλά όχι σε όλες. Οπότε τι γίνεται με την επιστροφή των δαπανών. Και το θέμα των ομοιόμορφων εγγράφων για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία αυτών των ψηφιακών αντιγράφων των δεδομένων. Το ψήφισμα προτείνει ευκολότερη και ε, άμεση πρόσβαση των ασθενών με κάποια τεχνολογία πληροφορίας. Θα πρέπει όμως να καθορίσουμε αυτή την ε, ε, ψηφιακή διαδικασία, γιατί από τα στοιχεία της Ευρωστάτ προκύπτει ότι 57% των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν πολύ το Ιντερνετ είναι άνω των 60 ετών, 60 με 75 ετών. Αυτοί είναι όμω που χρειάζονται περισσότερο η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Πολωνία. Μόνο 22%, 22 ε, των πολιτών δεν χρησιμοποιεί καν το διαδίκτυο. Οπότε, όντω ε, ε, οι ασθενείς που θα έχουν πρόσβαση στα, στα ψηφιακά δεδομένα θα έχουν πρόσβαση και σε τέτοιες υπηρεσίες και προσοχή στην προστασία των δεδομένων. Ε, τι γίνεται σε περίπτωση πανδημίας και πώς θα εξασφαλίζεται η κοινή χρήση. Ε, υπάρχει λογική στην, ε, στις προτάσεις αυτές. Επίσης έχουμε πολύ σοβαρή μεταναστευτική κρίση. Στην περίπτωση ελέγχου των συνόρων, ποιος στα αεροδρόμια ή στα λιμάνια ή στα χερσαία σύνορα θα κάνει τον έλεγχο αυτών των δεδομένων. οι φορείς του ελεκτικού μηχανισμού τι πρόσβαση θα έχουν στα δεδομένα αυτά. Επίσης, ε, μιλούμε για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών. Εκεί προτείνουμε συγκέντρωση δεδομένων ε, σε πραγματική μορφή, ενώ ε, οι παγκόσμιες εταιρείε προτείνουν κάποιες λύσεις μέσω των έξυπνων τηλεφώνων ή του smartwatch. Ε, επίσης υπάρχουν ε, ε, εφαρμογές που ελέγχουν την πίεση, τους, καρ, τους παλμούς της καρδιάς. Μήπως όμως έτσι γίνει μια απόπειρα εξαγωγής ιατρικών στοιχείων, κάτι που παραβιάζει την ιδιωτικότητα του ασθενούς. Θα πρέπει να προσέξουμε μήπως κάποια ιατρικά ιστιτούτα ή άλλοι φορείς έχουν ανεξέλεγκτη και απεριόριστη πρόσβαση σε τέτοιου δεδομένα, κάτι που είναι απαράδεκτο. Αυτά και όλες αυτές τις ανησυχίες θα τις περιλάβω στις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρίς από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο τέλος του μήνα το Βέλγιο θα προτείνει την πλατφόρμα για τις εφαρμογές των συνδεδεμένων ε, μέσων που θα συμπληρώνει τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών και πολλές άλλες χώρες θα αναλάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίε. Κάτι που δείχνει πόσο κρίσιμο είναι το ψηφισμά μας και το έτοιμά μας να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να ε, παρακολουθήσουμε αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ε, για παράδειγμα, θα, έχουμε τακτική, θα μπορούμε να παρακολουθούμε τη, το γλυκαιμικό, το, τη γλυκαιμία ενός ασθενούς και να ξέρουμε πόσο, πότε χρειάζεται να λαμβάνει το φαρμακό του. Βέβαια, θα πρέπει να, να σεβαστούμε οπωσδήποτε κάποιες αρχές ε, της προστασίας των δεδομένων. Νομίζω ότι είναι πολύ ορθολογικές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά έχω εδώ τρία σχόλια. Θέλουμε με το ψήφισμά μας να μεριμνήσουμε ότι όλα τα επιγραμμικά συστήματα θα πληρούν αυστηρέ προδιαγραφές ασφάλειας των δικτύων και πληροφοριών. Εδώ θα είμαστε αδιάλακτοι, ανένδοτοι. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων των ασθενών, που είναι σαφώς προσωπικού χαρακτήρα. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ώστε να έχουμε ένα πραγματικό ε, πανευρωπαϊκό σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντα τη διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων και προτυποποίηση των μορφοτύπων. Και επίσης, ακρογωνίως λήθος όλη αυτή τη πρόταση είναι η εξασφάλιση, κάτι που δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμή, τη ε, διαβίου κατάρτιση και των ε, ε, ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, των φαρμακοποιών για θέματα της ψηφιακής, της ηλεκτρονικής υγείας. Γιατί βλέπουμε ότι ο πληθυσμός μας γυράσκει, οι ασθενείς ταυτόχρονα γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί ω προς την ποιότητα και την εξατομήκευση των υπηρεσιών ε, και της ατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης και αυτή η ψηφιακή επανάσταση μας δίνει τη δυνατότητα να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις, ε, στις υπηρεσίες ε, υγείας και στην περίθαλψη. Θα πρέπει όμως να καθορίσουμε τους κανόνες και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ψήφισμά μας. Thank you. And next from... Ευχαριστώ. Γκουε. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να στηρίξει την ε, ψηφιακή μεταρρύθμιση στην υγεία. Και βεβαίως πρέπει να συνεχιστεί και η κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού για να γίνει αυτό. Τα συζητήσαμε τα θέματα αυτά πριν από δύο χρόνια, όταν συζητήσαμε τις ιατρικές συσκευές. Και συζητήσαμε όλες τις πλευρές της ηλεκτρονικής υγείας, το e-health και το m-health. Τι έχει κάνει συγκεκριμένα ε, έκτοτε η Κομισιόν. Ξέρω δεν έχει κάνει αρκετά. Δεν μου αρέσει. Και μάλιστα είναι σκανδαλώδες ότι δήλωσε ότι οι ψηφιακές λύσεις ε, δεν προχωράνε αρκετά. Και μάλιστα ε, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος ε, είναι πολύ διαφορετικό το επίπεδο. Μα δεν είναι δυνατόν να λέω αυτά τα πράγματα. Είναι γελία. Νομίζω ότι ένας διευθυντής ενός μικρού νοσοκομείου σε μια μικρή μας πόλη θα μπορούσε να πει αυτά που μας λέτε εδώ πέρα μετά από μισή ώρα δουλειά. Δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση πώς θέλουμε όντως να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες στην ε, περίθαλψη. Δεν έχουμε κοινέ ευρωπαϊκές λύσεις για τα θέματα αυτά. Δεν υπάρχει ανταλλαγή των αποτελεσμάτων, ε, της έρευνας, οι βάσεις ε, δεδομένων δεν επικοινωνούν. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, επιδημιών ή σπανίων ασθενειών. Αν ανταλλάσσαμε σωστά πληροφορίε, αν είχαμε υπερβεί τον κατακαιρματισμό των συστημάτων Υγεία, θα είχε πολύ θετικό αντίκτυπο και οικονομικό. Γιατί όπως ξέρετε ζούμε σε μια εποχή όπου το ε, smartwatch σου μπορεί να μετρήσει <clears throat> τη, το, τους φυγμούς σου και να δώσει πληροφορίες, να τις στείλει απευθείας στο γιατρό σου. Σε μια τέτοια εποχή που ζούμε δεν μπορούμε ούτε καν να ε, ε, έχουμε πρόσβαση σε όλες μας τις ιατρικές εξετάσεις. Και ούτε ο γιατρός μας. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Και οι ορισμοί είναι ανεπαρκείς. Πώς θα ορίσουμε την ανάγκη της ή ε, τεκμηρίωσης. Σε ποιον ανήκει η τεκμηρίωση του ιστορικού του ασθενούς. Και πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχει επικάλυψη, για παράδειγμα, ε, ε Πηγαίνουμε σε διάφορου γιατρού και μα κάνουν την ίδια θεραπεία, γιατί κανεί δεν ξέρει τι έχει γίνει. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέσα. Βέβαια, ε, είναι το θέμα της κατάρτισης. Εάν αύριο τα, ε, ε βάζα, τα, άρχισαν να λειτουργούν όλα αυτά, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν γιατί ούτε οι γιατροί ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό δεν θα ήξεραν πώ να τα να χρησιμοποιήσουν γιατί έχει καθυστερήσει η κατάρτιση. Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένε Πολιτείε δείχνουν τον δρόμο. Ο πληθυσμό μα γερνάει όλο και περισσότερο. Είναι ζωτική σημασία να έχουμε αυτά τα εργαλεία. Αυτά που μα προτείνει η Κομισιόν δεν με πείθουν ότι θα υπάρξει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Και επίση υπάρχουν και περικοπέ ε, περικοπές στους ε, ιατρικούς προπολογισμού. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Στον τομέα αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα απασχολήσει και τη νέα Επιτροπή. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα γίνουν ολένα και πιο απαιτητικοί στο μέλλον στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής που επιθυμούν να τον λάβουν. Η κυρία Καμπεθόν Ρουίφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω την άποψή μου για το θέμα αυτό, διότι θεωρώ ότι η ψηφιακή υγεία είναι ένα θέμα όπου είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε ψηφιακά μέσα και στην υγειονομική περίθαλψη και να βελτιώσουμε την πρόσβαση των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως το θέμα είναι πιο λεπτό από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ιδιωτικότητα και τον ιδιωτικό βίο των ανθρώπων. Έχει να κάνει ε, με με το σύστημα υγείας συνολικά και το κατά πόσον είναι δίκαιη η πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Και επίσης σημαντικό είναι πως ασκεί κανείς το δικαίωμά του στην πρόσβαση στην ε, υγεία. Υπάρχουν ε, πολλά θέματα που σχετίζονται με αυτό, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει εδώ και μια διάσταση επιχειρηματική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση και αν δούμε τις τελευταίες ε, ανακοινώσει των τελευταίων ετών θα δούμε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν ε, εγκρίνει την πρόσβαση του οποιοδήποτε στα δεδομένα τους. Εδώ όμως θέλουμε υποτίθεται να βασιστούμε και στην αλληλεγγύη, δηλαδή τα περισσότερα συστήματα που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για τους ε, ανθρώπους που είναι ε, ασθενείς, τα περισσότερα κόστη καλύπτονται από τους υγιείς. Αυτό σημαίνει... Ότι μερικές φορές είναι τόσο ε, πολυδάπανη θεραπεία που τελικά όλη η κοινωνία καλείται να τη χρηματοδοτήσει. Αυτό είναι το νόημα των δαπανών της υγείας. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στην υγεία. Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε ασθενούς. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι τα εθνικά συστήματα υγείας και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποτελέσουν απαραίτητο κρίκο και σημαντική φωνή στη διαχείριση ε, των δεδομένων και στο θέμα της ψηφιακής υγείας. Γιατί αυτά τα στοιχεία έχουν οικονομικό ενδιαφέρον και μπορούν να επηρεάσουν το σύστημα υγείας ε, εφόσον χρησιμοποιηθούν από το σύστημα υγείας και τα υγειονομικά συστήματα είναι οι καλύτεροι θεματοφύλακες του ελέγχου ε, της χρήσης των δεδομένων και της, ε, του σεβασμού της ιδιωτικότητας των ασθενών. Οπότε θα πρέπει να επικεντρώσουμε τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση στα κράτη-μέλη και στα εθνικά συστήματα υγείας. Αυτά θα πρέπει να είναι τα αρμόδια για τη διαχείριση και τον έλεγχο της διαχείρισης των δεδομένων. Οπότε είναι η ευκαιρία, αλλά μην είμαστε αφελείς, γιατί το θέμα είναι πολύ λεπτό και ευαίσθητο και σε τελική ανάλυση μπορεί να επηρεάσει την δικαιοσύνη, την ισοτιμία, την ισότητα και την πρόσβαση του ασθενού στο σύστημα. Γιατί δεν θα πρέπει να αποκεφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Γιατί χάρη στα αισθήματα υγείας συγκεντρώθηκαν αυτά τα στοιχεία. Και σίγουρα το σύστημα υγείας έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει και δεν μπορούμε να το παραγωνίζουμε. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την ισοτιμία, τη δικαιοσύνη και την πρόσβαση στην υγεία ως αναπαλωτήριο και θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τις απόψεις της. Ο κύριος Μαρσέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας για τη συζήτηση και την προσοχή που δίνουν στην συνέχιση της πρότασης που υιοθετήθηκε ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ε, υγεία στην ψηφιακή αγορά. Σίγουρα ε, τα δεδομένα υγείας είναι το κλειδί στον ψηφιακό μετασχηματισμό και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και καλύτερα δεδομένα θα οδηγήσουν σε καλύτερη υγεία, καλύτερο βιωτικό επίπεδο και άρα είναι προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη. Φυσικά λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη και τη σημασία της διαλειτουργικότητας. Οι, σύστα, οι τονίζουν την ανάγκη εξασφάλισης ε, ε, των ηλεκτρονικών ε, ιατρικών, της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρικών ιατρικών αρχείων και διασυνοριακά και θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εξέλιξη ενός σημαντικού σχεδίου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη για τη θέσπιση υποδομών, ψηφιακών υποδομών υγεία, ώστε κάποιε συνόψεις του ιατρικού μητρώου και συνταγέ να κυκλοφορούν διασυνοριακά. Ήδη πιλωτικά γίνεται τέτοια ανταλλαγή συνταγών και ιατρικών μητρώων από τις αρχές του 2019, Απρίλιο του 2019 και πολλές χώρες ε, θα συμμετέχουν μέχρι τα τέλη του 2020. Όλες οι χώρες θα συμμετέχουν μέχρι τα τέλη του 2021. Δίνουμε έμφαση λοιπόν στη διαλειτουργικότητα και θα λάβουμε υπόψη ε, τις προτάσεις σας για τους μορφότυπους ανταλλαγή των ηλεκτρονικών ιατρικών μητρών. Αυτό θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της ε, διασυνοριακής πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα. Συμφωνούμε ότι η πρόσβαση των πολιτών στα στοιχεία υγείας τους θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο και με σεβασμό της αρχής ιδιωτικότητας και των κανόνων του Γενικού Κανονισμού προστασία των Δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει οι ψηφιακές υποδομές θα εδράζονται σε στιβαρά και ασφαλή πρωτόκολλα για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση Οπότε είναι σημαντικό το θέμα της ενημέρωσης και της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού και των ερευνητών. Η συνεργασία με τα κράτη-μέλη φυσικά θα έχει θεμελιώδη σημασία για την υλοποίηση των στόχων και χαιρετίζουμε τι συστάσει σας για ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στις αλλαγές ε, που θέλουμε, ώστε να γίνει ανθρωποκεντρική αυτή η ψηφιακή μετάβαση και σίγουρα ο μετασχηματισμός να λάβει υπόψη και την ανάγκη ένταξης ή έλλειψη αποκλεισμών στην ψηφιακή ε, αγορά. Και φυσικά θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τα απαραίτητε ε, τις δεξιότητες για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το ψηφιακό μετασχηματισμό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Um, the timetable... Λοιπόν, προθεσμία για τροπολογίες 16 Δεκάτου 11 ώρα το πρωί θα ψηφίσουμε στην ΕΝΒΗ 26-27 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Και τώρα, το επόμενο θέμα. τα συμπληρωματικά ε, ε, ε, πιστοποιητικά προστασίας για τα φάρμακα. Τίμο Βέλκεν, ο 4 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια πρόταση για αλλαγή του κανονισμού για το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα. Το Κοινοβούλιο, εδώ και αρκετό χρόνο, έχει ζητήσει μια εξαίρεση για την κατασκευή. Αυτό έχει να κάνει με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά από το Μάιο του 2016 και για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα. Αυτό το αναφέρουμε και στην αιτιολογική σκέψη. Όταν μπήκε αυτό το, εισήχθη αυτό το πιστοποιητικό για πρώτη φορά, ήθελαμε να δώσουμε κίνητρα για να υπάρχει έρευνα για καινοτόμα φάρμακα και λειτουργήσε πολύ καλά στη Δανία για παράδειγμα. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εκεί γενώσιμη ε, φαρμακοβιομηχανία και επίσης και καινοτόμα. Αλλά ο κόσμος αλλάζει. Και τώρα βλέπουμε ότι η παραγωγή των βιομοειδών και γενοσύμων στην Ένωση έχουν ένα πρόβλημα ανταγωνισμού. Δηλαδή, οι φαρμακοβιομηχανίες εκτός της Ένωσης έχουν πλεονέκτημα. Πρέπει λοιπόν να καταργηθεί. Με την τροπολογία του κανονισμού αυτού θέλουμε να υπάρξει ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών εντός και εκτός της Ένωσης. Και χαιρετίζω λοιπόν αυτό το στόχο. Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των δικών μας φαρμακοβιομηχανιών, ιδιαίτερα για να μπορούν να κάνουν και εξαγωγές, εκεί που δεν υπάρχουν τέτοια πιστοποιητικά, κάνουμε ένα σωστό βήμα. Και φυσικά διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να προστατεύουμε την ε, πνευματική διοκτησία. Γι' αυτό προβλέπω πέντε χρόνια. Και δεν προτείνω στην γνωμοδότησή μου ακριβώς καμία αλλαγή αυτής της προθεσμίας. Η αλλαγή του κανονισμού όμως έχει και μία άλλη πλευρά αυξάνεται η προσβασιμότητα των πολιτών μας ε, στα φάρμακα γιατί τα, οι τιμές των νέων φαρμάκων αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες τόσο πολύ που ορισμένες φορές δεν μπορούν να τα πληρώσουν πολλοί πολίτες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μειωθούν τα φάρμακα, ε, συγγνώμη, να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων μέσω χρήση περισσότερων γενοσύμων και βιομοειδών και για να έχουμε τη δυνατότητα ε, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα φάρμακα από την πρώτη μέρα, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο τις ε, εξαγωγές αυτές εξαιρέσεις, αλλά και την αποθήκευση αυτών των φαρμάκων. Έτσι βοηθάμε τους παραγωγούς μας εντός της Ένωσης και δεν θα έχουν κανένα κίνητρο να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε τρίτες χώρες. Και έτσι θα γίνουμε κέντρο φαρμακευτικής καινοτομίας και ιδίω για τον τομέα των βίο-ομοιδών Δεν είναι δυνατόν σε έναν τόσο σημαντικό τομέα να μεταφέρεται η παραγωγή στις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία. Συνοψίζοντας, γι' αυτό προτείνω στη γνωμοδότησή μου περισσότερα μέτρα ασφαλεία με βάση την οδηγία για τα παραποιημένα φάρμακα, να υπάρχουν διορθωτικοί μηχανισμοί που να μην είναι χαλαροί και να υπάρξουν εξαιρέσεις για τους ε, ε, κατασκευαστές, για τους φαρμακοβιομήχανους, για τις φαρμακοβιομηχανίες, για να μπορούν να αξιοποιούν αυτά τα φάρμακα την πρώτη μέρα. Και επιπλέον, η δυνατότητα να υπάρχει αποθήκευση δεν θα πρέπει να εμποδιστεί λόγω της υποτιθέμενης παραβίασης κανόνων εμπορικής πολιτικής. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία τέτοια σκέψη και δεν έχω ακούσει καμία τέτοια αντίρρηση. Η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης 16 Δεκεμβρίου. Και ε, θα το συζητήσουμε με του αδέλφους. Ευχαριστώ πολύ για το ΕΛΚ. Ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Λοιπόν, κοιτάξτε, ποιο είναι το βασικό με το οποίο θέλω να αρχίσω. Έχουμε πολύ ισχυρή προθεσμία για τις φαρμακοβιομηχανίες μας. Γιατί χρειάζονται για να μπορέσουν να αναπτύξουν νέα φάρμακα γιατί είναι περίπλοκη και δαπανήρια αυτή η διαδικασία. Εμείς θέλουμε να μπορούν να επενδύσουν σε νέα φάρμακα. Χρειαζόμαστε ισχυρή διανοητική ιδιοκτησία. Γιατί μόνο έτσι καλύπτονται οι κίνδυνοι. Και δεν είναι μόνο θέμα επενδύσεων και απασχόλησης. είναι η δυνατότητα να θεραπεύουμε ασθένειε. Άρα θέμα ζωή και θανάτου. Όχι μόνο για του συμπολίτε μα, αλλά παντού για του ανθρώπου στον κόσμο. Από αυτή την οπτική γωνία πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτή η πρόταση υπονομεύει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Δεν νομίζω ότι είναι ε, η σωστή προσέγγιση. Και στέλνουμε λάθο μήνυμα αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και θέλω να το πω για να το ξέρετε όλοι. Αλλά αφού έχει υποβληθεί αυτή η πρόταση. Ε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Άρα κυρίως να ασχοληθούμε με την ε, εφαρμογή, να εφαρμοστεί σωστά. για να μην ε, υπονομεύσει και άλλα τμήματα του πλαισίου πνευματικής διοκτησίας. Τώρα για αυτή τη γνωμοδότηση που συζητάμε τώρα εδώ. Όχι την ίδια την πρόταση, τη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι είναι αρκετά αντικειμενική. Και χαίρομαι που το διαπιστώνω. Έχει πολύ καλά στοιχεία και δεν περιέχει, και αυτό είναι πιο σημαντικό, κάτι που πολύ θα με ανησυχούσε εάν είχε συμπεριληφθεί. Καλό είναι που δεν ζητάει και αναδρομικότητα ο κύριο Βόλκεν. Πρέπει από κοινού να απορρίψουμε την αναδρομικότητα, γιατί αν κάναμε κάτι τέτοιο, τότε στην ουσία θα καταργούσαμε τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. και θα είχαμε και νομικά προβλήματα. Καλό λοιπόν που δεν έχουμε τέτοια αναδρομικότητα. Νομίζω ότι ε, σωστά είναι και τα μέτρα για την εξαγωγή σε χώρες που δεν έχουν τέτοια συμπληρωματικά πιστοποιητικά. Καλό αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τίποτα δεν είναι τέλειο. Υπάρχουν δύο θέματα όπου διαφωνώ για αυτή, σε αυτή τη γνωμοδότηση, με αυτή τη γνωμοδότηση. Και πιστεύω ότι πρέπει να τα δούμε για να διατηρηθεί η διανοητική διοκτησία. Και το πρώτο είναι, λυπάμαι γιατί έχω ακούσει, είναι το θέμα της αποθήκευσης. Δεν νομίζω ότι ο κανονισμός θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει την αποθήκευση. Γιατί μειώνεται η πρόσβαση στα γενώσιμα. Δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι και η Επιτροπή ήδη λένε στην πρότασή της ότι μία φαρμακοβιομηχανία που ήδη εξάγει θα μπορούσε να μπορεί να ε, παράγει και για την ενιαία αγορά όταν θα λύγει αυτό το συμπληρωματικό πιστοποιητικό. Υπάρχει ανάγκη, θα αλλάξει ο ουσιοδός κατάσταση, αν μπορεί να αποθηκεύσει κάποια τέτοια. μελέτησα και διάφορες, ε, διάφορα κείμενα από αυτού που λένε ότι είναι τόσο πολλοί άλλοι παράγοντες που αφορούν τη διάθεση στην αγορά. Όχι απλώς η αποθήκευση. Παράγοντες λοιπόν που δεν επηρεάζονται καθόλου από την αποθήκευση. Γιατί θέλει η γνωμοδότησή σας να αποδυναμώσει την πρόταση τη Επιτροπής όσον αφορά την ε, γνωστοποίηση. Θα πρέπει να ε, γνωστοποιείται ο κάτοχος του πιστοποιητικού. Θα πρέπει να μπορέσει ο καθένας να δει αν ο παραγωγός του γενώσιμου ε, συμμορφούνται με τις προδιαγραφές. Είναι ουσιώδες. Αν θέλεις ο κάτοχος του πιστοποιητικού να δει εάν το προϊόν υπάρχει σε αυτή τη χώρα ούτως ώστε ο κάτοχος του πιστοποιητικού να ε, μπορεί να δράσει γνωρίζοντας την κατάσταση όσον αφορά τον ανταγωνισμό και βεβαίως η πληροφόρηση αυτή θα είναι εμπιστευτική και επιπλέον και πολύ σημαντικό. Ερώτηση προς την Επιτροπή. Είμαι μέλος τα τελευταία 14 χρόνια της ΙΝΤΑ και αυτό το πιστοποιητικό SPC είναι θέμα που το είχαμε σε πολλές διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Και αν το συζητήσουμε τώρα με αυτούς που διαπραγματεύονται εμπορικές συμφωνίες, βεβαίως ακόμη πολλοί ζητάνε τέτοια πιστοποιητικά. Το επιβάλαμε, όχι δεν το επιβάλαμε, το ζητήσαμε και το δέχτη ο Καναδάς. Αυτό δεν αποδυναμώνει τη δυνατότητά μας να ζητήσουμε να συμπεριλαμβάνονται αυτά τα SPC διαπραγματεύσεις και θα ήταν συμβατό με τι επάρχουσε συμφωνίες μας ελευθερου εμπορίου. Αυτό θέλω να ρωτήσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίω. Μ' αρέσει όπω είπα το σχέδιο γνωμοδότησή σα παρά το ότι διαφωνώ σε κάποια σημεία και βεβαίω θα συνεργαστούμε μαζί. Επόμενο από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, η κυρία Κρούπα. Θα ζητήσω από όλου να παραμένουν στο τετράλεπτο. Ευχαριστώ. Η παρασκευή γενώσιμων και βιομοειδών φαρμάκων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ε, υπόκειται σε συγκεκριμένε και πολύ πιο αυστηρέ προδιαγραφέ από ό,τι στην Παρασκευή εκτό Ένωση. Γι' αυτό και η πρόταση επιλύει κάποια προβλήματα για του κοινοτικού παρασκευαστέ φαρμάκων, γενώσιμων και βιομοειδών. Καλό το σχέδιο γνωμοδότηση. Δεν καταστρατηγεί κανένα καμία διάταξη της οδηγίας ούτε κανονισμού διευκολύνει απλώς την πρόσβαση ε, σε γενώσιμα φάρμακα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και δυνατότητα να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Και από ιατρική σκοπιά θα ήθελα να πω ότι κάθε αλλαγή από το πρωτότυπο σε γενώσιμο φάρμακο μπορεί, θα, και θα πρέπει να συνδυάζεται με την ανάγκη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Και ναι, μεν θα πρέπει να γίνονται έρευνε για την ασφάλεια του φάρμακου, αλλά μερικέ φορέ είναι τόσο δαπανηρέ αυτέ οι έρευνε και γίνονται τόσο ακριβά αυτά τα φάρμακα, ιδιαίτερα από ε, μία περίοδο και μετά, που έχει νόημα αυτή η πρόταση. Και φυσικά ε, να προσέξουμε για να μην γίνεται παραποίηση η νοθεία αυτών των γεννόσιμων φαρμάκων. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, and Ευχαριστώ. Α, όχι, έφυγε. Λοιπόν, υπάρχουν άλλα μέλη της Επιτροπής που θα ήθελαν να συμβάλλουν. Καμπεθόν Ρουίθ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επενέσω τον συνάδελφο Βέλκεν για την αξιόλογη προσπάθειά του και την καλή του πρόταση που είναι ισορροπημένη και σωστή. Άρτια. εγώ δεν έχω διαφωνίες ε, με τον εισηγητή. Απλώς θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Το γεγονός ότι επιτρέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που εκπνέει η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Άρα δεν ισχύει πια το πνευματικό δικαίωμα. Από τη στιγμή που ε, εισέρχεται αυτό το προϊόν στην ε, εσωτερική αγορά και τα γενώσιμα που παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα βελτιώσει την κατάσταση της, ε, του ανεφοδιασμού με σε φάρμακα και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Θα στηρίξει τα συστήματα υγείας που καθυστερούν περίπου ένα εξάμεινο ε, για να εισάγουν πλήρως τα γενώσιμα από τη στιγμή της Παρασκευής του μετά την εκπνοή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε επίσης την πρόσβαση των ασθενών στα γενώσιμα φάρμακα και αυτό το καταφέρουμε χάρη στην ε, πρόταση και θα βελτιώσουμε και την απασχόληση σε ένα κλάδο που χρειάζεται επίσης ανταγωνιστικότητα. Εγώ βλέπω σημαντικές ευκαιρίες με την πρόταση αυτή. Και αν εμείς δεν παράγουμε εντός τη Ευρωπαϊκής Ένωση πρώτα, θα χρειαστεί να εισάγουμε. Δηλαδή θα αγοράζουμε από τρίτε χώρε. Ενώ θα μπορούμε ταυτόχρονα να παρασκευάζουμε εδώ τα φάρμακά μα. Απαράδεκτο. Και σίγουρα δεν επηρεάζεται η πνευματική ιδιοκτησία, γιατί αν υπήρχε πρόβλημα πνευματική ιδιοκτησία, κανονικά θα έπρεπε να εισάγουμε καν. Δεν είναι θέμα πνευματική ιδιοκτησία. Εδώ. Υπάρχει μια ανομαλία στην ερμηνεία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει μια στρέβλωση. Και ε, αυτή την ανομαλία κατοχυρώνει ο κανονισμός. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία αυτή η πρόταση. Επίσης, ε, για την κοινοποίηση θα είχε νόημα αν απαιτούσαμε και από τι εισαγωγή το ίδιο. Γιατί να αποχρεώνουμε σε κοινοποίηση τι τις δικές μας επιχειρήσεις και να απαλλάσσουμε τους, ε, τις τρίτες χώρες, τους παρασκευαστές τρίτων χωρών αυτό φέρει σε δυσμενή θέση τους δικούς μας παρασκευαστές και σίγουρα ο αρμόδιος κανονισμός, ο ρυθμιστικός ε, φορέας, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει την κοινοποίηση. Και αυτό να ισχύει και σε άλλους τομείς. Το να επιβάλλουμε ουσιαστικά τόσα κριτήρια σε επιχειρήσεις ώστε να τις αποτρέπουμε να παρασκευάσουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτο. Και ναι με κοινοποίηση αλλά ισορροπημένη και όχι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας του κλάδου χωρίς να υπονομεύουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Είναι καλή πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη βελτίωσε ακόμη περισσότερο ο κ. Βέλκερ. Θα πρέπει να αποφύγουμε τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων και να επιτρέψουμε στη φαρμακοβιομηχανία μα να παρασκευάζει εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργεί αποθέματα και από την πρώτη μέρα εκπνοή του διπλώματο ευρυστεχνία να μπορεί να τα διαθέτει στην ευρωπαϊκή αγορά. Ευχαριστούμε κ. Πέτερλε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Όταν μιλάμε για το να επιτρέψουμε στους ε, ευρωπαίους παραγωγούς γενοσύμων και άλλων βιοφαρμάκων να ανταγωνίζονται. Δεν σκεφτόμαστε πάνω απ' όλα τις εταιρείες και τα κέρδη τους, αλλά τους ασθενείς και το πώς μπορούν έγκαιρα να παίρνουν τα φαρμακά τους. Η σύντομη, η έγκαιρη παραγωγή των ε, γενώσιμων και των ε, βιο, αντιστοίχων, βιολογικά αντιστοίχων φαρμάκων τους, των δύο ομοειδών είναι κάτι που θα πρέπει να υποστηριχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν υπάρχει παραβίαση των συμβάσεων και των ε, ε, ε, αδειών μέχρι την τελευταία μέρα παρουσίας του στην αγορά. Θα πρέπει η ίδια η παραγωγή, η σύνθεση και η Παρασκευή να οδηγεί στην άμεση θέση στην αγορά των φαρμάκων μόλις λήξουν οι άδειε χωρίς οι παραγωγοί που έχουν εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθούν σε χειρότερη θέση από αυτούς που βρίσκονται εκτός Ένωσης. Είναι προς, δικό, προς το δικό μας ευρωπαϊκό συμφέρον όσοι παράγουν γενώσιμα και βιομοειδή ε, να παραμένουν στην Ένωση και όχι να πάνε σε τέτοιες χώρες. Ευχαριστούμε κυρία Γκροστέτ. Έψαχνα το κουμπί μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα γενώσιμα και τα δύο πρέπει να θεωρηθούν ε, στυλοβάτες της ε, ιατρικής αγοράς των φαρμάκων, προφανώς. Όμως σημαντικό είναι να μην αναπτυχθούν τα μένεις βάρος των δε, διότι πρέπει να παραμείνει η ανάπτυξη, η καινοτομία και η έρευνα εδώ. Διότι το βιομοειδές του σήμερα είναι το γεννόσιμο το αύριο. Δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε και το σύστημα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά να δούμε και με θετικό μάτι τα γεννόσιμα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει την παρασκευή γενώσιμων φαρμάκων στην Ευρώπη πριν την εκπνοή των αδειών για τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων φαρμάκων. Μόνο για την εξαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όντω πάει στη σωστή κατεύθυνση για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παραγωγών γενοσύμων και βιομοειδών. Του επιτρέπουμε να παίξουν ε, το σωστό ρόλο, ε, να παίξουν μάλλον ε, με ίδιους κανόνες το παιχνίδι του ανταγωνισμού με τους αντιπάλους τους. Τώρα για την αποθήκευση και σε σχέση με αυτά που λέει ο εισηγητής μου φαίνεται σημαντικό τα γενώσιμα και τα δύο όμοειδή να ενισχυθούν περισσότερο, να παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε τρίτες χώρες, είναι σημαντικό, αλλά επίσης βάσιμο είναι το επιχείρημα για τους ε, παραγωγούς των καινοτόμων φαρμάκων, των νέων φαρμάκων το να θέσουμε ένα αμφιβόλο το, το πλαίσιο παρότρεξης προς την καινοτομία δεν θα ενθαρρύνει τους καινοτόμους να ασχοληθούν με την ανάπτυξη και την έρευνα. Θα πάνε σε χώρες όπου το νομικό πλαίσιο είναι ευνοϊκότερο ε, προς την προστασία της πραγματικής ιδιοκτησίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν νομίζω θα ασφάλουμε εάν επιμείνουμε. Ε, εάν ένα τέτοιο μέτρο ε, δεν κατέφερε ένα κέριο πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα, θα ήταν παρόλα αυτά ένα αρνητικό μήνυμα ε, εις βάρος της εμπιστοσύνης, εμπιστοσύνης που είναι απαραίτητη για να τονώσουμε τις επενδύσεις με προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζω ότι είναι σημαντικό για τα υγειονομικά μας συστήματα να βελτιώσουν τη δίσδυση στην αγορά των γενοσύμων και ομοειδών, δύο ομοειδών, όμως νομίζω ότι πρέπει να επιφυλαχθούμε να προβλέψουμε την αποθήκευση ως εξαίρεση ε, ως λύση και ως λύση θαύμα. Ε, θα πρέπει εγκαίρως να φτάνουν τα γενώσιμα στην αγορά και να μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η ανάγκη εξαίρεση στην αποθήκευση είναι κάτι που θα μπορούσε να κρυθεί ε, μεταγενέστερα, κάτι που ίσως να είναι όντω επικοδομητικό. Είμαι βέβαιη ότι ε, μπορούμε να κάνουμε και άλλε βελτιώσει στο κείμενο τη Επιτροπή για να βεβαιωθούμε ότι οι στόχοι τη ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα παραγωγή γενοσύμων και γίνεται σεβαστό και αυτό θα κάνω και εγώ η ίδια υποβάλλοντα μια σειρά από τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα λόγω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Φερχούβεν. Ευχαριστώ πολύ. Μερικά σχόλια για όσα άκουσα ως τώρα. Με χαρά άκουσα ότι υπάρχει ευρεία συνένεση, ότι η πρόταση είναι επικοδομητική και εξισορροπημένη. Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω εργασία. Μερικά σχόλια για τις δηλώσεις που έγιναν. Το θέμα της αποθήκευσης. Όπως εξηγήσαμε στη μελέτη τύπου κατά την άποψή μας δεν χρειαζόμαστε την αποθήκευση καθόλου. για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Αν δείτε τη μελέτη αντικτύπου, τα περισσότερα οικονομικά ωφέλη που επιδιώκουμε με την πρόταση αυτή, κέρδος από τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και αν στην Ευρώπη, έχουν να κάνουν με την ε, εξαγωγή, όχι με την αποθήκευση. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο ευρώ παραπάνω το χρόνο. Είναι τεράστιο το ποσό. Κοιτάξτε τις ε, μελέτες η αποθήκευση αυτή καθεαυτή δεν προσθέτει και πολλά. Είδαμε τα προβλεπόμενα ωφέλη, κάναμε μια μέτρηση και είδαμε ότι είναι ελάχιστα και υπάρχει βέβαια πάντα το πρόβλημα της πρόσβασης στα φάρμακα. Εάν αυτό επιληθεί, Ε, αρκεί η εξαίρεση για τις εξαγωγές και τότε λύνουμε ένα μεγάλο πρόβλημα για την παραγωγή. Εάν δούμε λοιπόν την οικονομική ανάλυση εδώ, βλέπουμε ότι η αποθήκευση απλώς δεν είναι απαραίτητη. Και επίσης να πω ότι η πρόσβαση στα φάρμακα προφανώς είναι πολύ σημαντική, αλλά η πρότασή μας δεν μπορεί να πάει παραπέρα ως προς αυτό. Ε, υπάρχει και μια γενικότερη συζήτηση για την οποία είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίε. Θα ασχοληθεί με την πρόταση για τα σχετικά κίνητρα. Αλλά α μην ε, φορτώσουμε πάρα πολύ αυτή την πρόταση με όλα τα θέματα τη πρόσβαση στα φάρμακα τώρα ω προ τον ενιαίο ταυτοποιητή. Όπω ξέρετε, αυτό ο ενιαίο ταυτοποιητή έχει προωθηθεί από την ε, οδηγία των οθευμένων φαρμάκων. Το εισάγαμε ως μέτρο ε, για να βελτιώσουμε την υγεία και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και αυτή είναι και η πρόθεση αυτής της ε, νομοθετικής πράξης. Ξέρουμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ξέρουμε ότι και σε αυτό το νομοθέτημα πρέπει να προβλέψουμε αυστηρέ προποθέσει για τον ενιαίο ταυτοποιητή. Όμως εδώ μιλάμε για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι γενικώ πρόθεση τη υγεία και τη ασφάλεια στην Ευρώπη το πρόβλημά μα. Σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε κοινοποίηση, να εξηγήσω ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει ως εξής. Προσπαθήσαμε να επιδιώξουμε ένα διτό στόχο. Η προσέγγιση μας θέλαμε να είναι ισόρροπη. Θεωρούμε ότι η διαδικασία κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να υπάρχει διαφάνεια και να προστατεύσουμε τα ε, δικαιώματα των κατόχων, των παραγωγών. Και θα πρέπει τα γενώσιμα και τα βιομοειδή να παράγονται με τρόπο που να υπάρχει ο μέγιστος δυνατός βαθμός διαφάνειας. Όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει και ε, η διάχυση και η διάδοση των απόλυτων πληροφοριών για τον ίδιο σκοπό. Γι' αυτό ε, ε, άκουσα ότι πρέπει να γίνουν προτάσεις για να αλλάξει αυτό το σήμα στο κείμενο και ευχαρίστω να τις δούμε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι η σωστή επιλογή. Ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα του κυρίου Φιέλνερ, εάν αυτό θέλουμε να κάνουμε με το waiver με την εξαίρεση. Ε, και αν αυτό συνάδει με τι διεθνεί μα επιχρεώσει. Θα έλεγα πω ναι, και το λέμε και ξεκάθαρα σε αιτιολογικέ σκέψη τη έκθεση. Αυτό που κάνουμε σήμερα συμπληρώνει τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτέ τι υποχρεώσει που προκύπτουν από τι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Διότι η πρόταση αυτή διατηρεί ένα σύστημα ε, δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. Ε, που είναι το σχεδόντερο στον κόσμο, συνεχίζει όμω να πουλάει και σε τρίτε χώρε. Αυτό κάνουμε. Το κάνουμε και επιτυχώ μάλιστα, όπω τα ξέρουμε, σε αυτό το πλαίσιο. Οπότε η πρότασή μα αυτή συμβαδίζει απολύτω με την προσέγγιση μα για τι ε, συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Νομίζω ότι μπορώ να πάψω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ξαναδώσω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Βέλκεν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους αδέλφους για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εντάξει, δεν εκπλήσει το ότι σε ορισμένα σημεία έχουμε διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στην ίδια την μελέτη αντικτύπου η Κομισιόν λέει ότι οι εξαιρέσει και για την παραγωγή και για την αποθήκευση και δημιουργία αποθεμάτων θα βοηθήσει να επιληθούν τα προβλήματα. Άρα η Διακομισιόν αναγνωρίζει ότι τα αποθέματα βοηθούν τους πολίτες. Τι έγινε το 2000 ενώπιον του ΠΟΕ. Κοιτάξτε, εκείνη την εποχή δεν, δεν είχαμε ακόμη SMS. Άρα ε, ο κόσμος έχει αλλάξει. Αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε όταν ε, παρουσιάζουμε επιχειρήματα. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η πρόταση αυτή ε, δεν αποδυναμώνει τα πνευματικά δικαιώματα. Και θεωρώ ότι με τα αποθέματα δεν θα επιτρεπόταν απλώς να πουληθούν όλα από κοινού. Είμαστε σε μια κοινότητα δικαίου, άρα να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε παρανομία μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε όντω θα προκύψει στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που θα υπάρξουν πολλές τροπολογίες ούτως ώστε να ε, βελτιώσουμε την περίθαλψη των συμπολιτών μας και ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος προθεσμία για τροπολογίες 16 Δεκάτου 11 το πρωί και θα ψηφίσουμε στην ΕΝΒΗ 26 και 27 Νοεμβρίου και στην Τζούρι αναμένεται να ψηφιστεί το θέμα αυτό τον Ιανουάριο του 19 και η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου 9 με 1. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι.